ladies and gentlemen, I think we can start. Να ξεκινήσουμε κυρίε και κύριοι και όσοι βρίσκεστε πίσω όρθιοι μπορείτε να περάσετε μπροστά και να κάτσετε. Θα ακούτε και την τερμηνία με τον τρόπο αυτό και θα έχετε και μικρόφωνο. Περάστε, περάστε και καθίστε μπροστά. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σα καλωσορίζω Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω και μία ομάδα από το Μέκλεμουρκ Φόμπορμεν, τα χαρή και ο φίλος μας ο Κούν. Σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή μας λοιπόν. Ίσως ε, όσοι κάθεστε παρακαλώ στέκεστε πίσω όρθιοι, μπορείτε να περάσετε μπροστά για να καθίσετε. Wir Καλώς ορίσατε λοιπόν στην ακρόαση για την ε, συμβολή ε, των ε, συστημάτων μεταφορών στους στόχους της Ευρώπης 2030 για την ενέργεια και το κλίμα. Ξέρετε ότι στο τέλη του μήνα έχουμε το μεγάλο, τη μεγάλη εκδήλωση το COP21 στο Παρίσι και γι' αυτό λοιπόν διοργανώσαμε και τη σημερινή ακρόαση. Χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε εδώ τόσου πολλού συμμετέχοντε και θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχά στον κύριο Τζιλ Παγνιό, ο οποίο και είναι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, ΕΝΔΙ και εισηγητή ε, τη έκταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ μια συμφωνία στο Παρίσι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου ζητήσατε να πάρω το λόγο σήμερα εδώ. Σας χαιρετώ όλους και όλους και χαίρομαι, ε, όλους και όλες και χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, που ξαναβλέπω μεταξύ άλλων τον Ντομινίκ Ρίκε, μαζί με τον οποίο ε, ε, έχω υπάρξει μέλος στην Επιτροπή Μεταφορών για πέντε ολόκληρα χρόνια, μεταξύ 2009-2014. Σήμερα αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το Περιβάλλον και την υγεία και τη διατροφική ασφάλεια. Είμαι μέλος και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αλλά και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχω την τιμή να είμαι ο εισηγητής ε, για αυτό το κείμενο ίδιας πρωτοβουλίας. Πρόκειται για μια νέα συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι και το κοινοβουλευτικό κείμενο ψηφίστηκε στις 14 του περασμένου Οκτωβρίου με ευρία πλειοψηφία πολύ μεγάλη πλειοψηφία ε, ε, και έτσι εγκρίθηκε η έκθεσή μου και οριστικοποιήθηκε η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διάσκεψη των μερών για το κλίμα 21 στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου στο Παρίσι. Και μάλιστα και, άλλοι, ε, και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την καθοδήγηση του Προέδρου Κανιέτε θα είμαστε παρόντες σε αυτή τη ε, μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι, όπου και θα υπερασπιστούμε προφανέστατα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τις δικές μας θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα μεταφορών. Κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις καταρχάς. Πρόκειται για τον αγώνα του αιώνα ε, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βεβαίως και πέρα από αυτή τη μάχη τα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να πούμε και το εξής. Εάν τίποτα δεν γίνει θα αυξηθεί παγκοσμίως η θερμοκρασία του πλανήτη κατά 4,5 έως και 6 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες θα γίνουν αμέσως αισθητέ από αυτή την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Για παράδειγμα να σας πω ότι στην επικαιρότητα ο τύπος και ο βέλγικος τύπος μεταξύ άλλων πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα βυθιστεί η πρωτεύουσα του Ομόσπονδου κρατηδίου του Βελγίου. Θα βυθιστούν οι Βρυξέλλες εάν αυξηθεί ε, η θερμοκρασία στον πλανήτη κατά 4,5 έως 6 βαθμούς μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Είναι μια ευκαιρία να βρεθεί λύση στο Παρίσι στην 21η διάσκεψη των μερών στο πλαίσιο των Ηνωμένων για το κλίμα όλοι παρακολουθούν αυτή την κινητοποίηση έτσι ώστε η Σύνοδος των Παρισίων να στεφθεί με επιτυχία ακόμα και οι χώρες που δεν θέλησαν να υπογράψουν το πρωτόκολλο του Κιώτο όπως ήταν η ΙΠΑ και η Κίνα εκείνη την εποχή γιατί μόνο 38 βιομηχανικές εκβιομηχανισμένες χώρες είχαν υπογράψει ε, τη συμφωνία Κιώτο το 1997. Σήμερα 150 χώρες έχουν ήδη υποβάλει την εθνική τους ε, συμμετοχή, την εθνική τους συνεισφορά και έτσι όπως έχουν οι συνεισφορές των κρατών μελών Έχουμε ήδη ε, καταφέρει να μειώσουμε αυτούς τους βαθμούς και θα αυξηθεί ε, η θερμοκρασία και το, στον πλανήτη μας κατά 2,7 βαθμούς και όχι 4,5 ως 6. Παρόλα αυτά εμείς θέλουμε στο Παρίσι να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει ε, την άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς maximum, το μέγιστο και όχι παραπάνω. Το διακύβευμα είναι τεράστιο όπως αντιλαμβάνεστε και πράγματι θέλουμε μια συμφωνία συνολική και είμαστε σε καλό δρόμο γιατί πάρα πολλές χώρες έχουν υποβάλει εθνικές προτάσεις και η ΙΠΑ και η Κίνα και άλλες χώρες, Νέα Ζηλανδία μεταξύ άλλων, είναι έτοιμες να συμβάλλουν. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ε, υπέγραψε μια πολύ σημαντική συμφωνία μαζί με τον ε, πρόεδρο της Κίνας. Πέρα λοιπόν από αυτή την συνολική οικουμενική συμφωνία, το σημαντικό είναι να έχουμε και μια συμφωνία που να είναι νομικός δεσμευτική, διότι το γνωρίζουμε οι καλές προθέσεις στα τέλη του 2015 μπορούν να αλλάξουν τελείως πρόσωπο και να ε, μεταφραστούν σε κάτι το τελείως διαφορετικό τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό εμείς θέλουμε να υπάρξει μια ρήτρα αναθεώρησης κάθε πέντε χρόνια έτσι ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της εθνικής συνεισφοράς, να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της εφαρμογής, της συμφωνίας των Παρισίων, έτσι ώστε κάθε χώρα να είναι νομικώς δεσμευ... δεσμευμένη να επανεξετάσει την πορεία της και την πρόοδό της αναλόγως και σύμφωνα με αυτό που θα έχει ήδη υπογράψει ε, κατά την έκβαση της 21ης διάσκεψης των μερών στο Παρίσι. Σαφέστατα είναι φιλόδοξη η στόχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων ε, μέχρι το 2030 ε, στην Ευρώπη κατά 25% Όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεσή μου και θα το πετύχουμε μόνο εάν ο κλάδος των μεταφορών συμβάλλει τα μάλα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Γιατί είναι ο δεύτερος κλάδος που εκπέμπει περισσότερα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου παγκοσμίω και τα συγκεκριμένα αέρια το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνονται η εκπομπή τους δηλαδή κατά 30% τα τελευταία 25 χρόνια. Πρέπει να ε, κάνουμε ε, το παν για να μειώσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, να το μετριάσουμε και έχουμε πέντε προτάσεις για το κλάδο των μεταφορών, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για τη μείωση των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Θα μπορούσαμε μέχρι το 2030 να έχουμε 30% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε ο κλάδος των μεταφορών ε, καταναλώνει ε, ευθύνεται για το 31,6% των εκπομπών αερίων σύμφωνα με την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο κλάδο των μεταφορών με την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, με τη γενίκευση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της χρήσης υβριδικών αυτοκινήτων, και ε, σε μεσοπρόθεσμη βάση με την ανάπτυξη πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θα πρέπει μέχρι το 2020 να καταργήσουμε πλήρως τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Σύμφωνα με ε, το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 4,5%. 5 δις έχουν κινητοποιηθεί ε, ως επιδοτήσεις στην εξόριξη ορυκτών καυσίμων. Από την Κίνα, από τη Ρωσία, από τη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα 700 εκατομμύρια δολάρια, από την Ιαπωνία 157 εκατομμύρια δολάρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, δίδονται τεράστιες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, καταργώντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, απελευθερώνουμε πάρα πολλά κονδύλια τα οποία μπορούμε να διοχετεύσουμε στις καθαρές πηγές ενέργειας έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτές και στις μεταφορές μεταξύ άλλων. Και θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι το στόχο των δύο βαθμών. Είναι αδύρυτη η ανάγκη για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής για την αλλιευτική δραστηριότητα θα πρέπει να κινητοποιηθούν για να μειωθούν οι εκπομπές και σε αυτούς τους κλάδους της οικονομίας. Στην έκθεσή μου δίνω έμφαση ε, και υποβάλλω συγκεκριμένες προτάσεις για το τομέα των εναέριων μεταφορών έτσι ώστε την Ευρώπη να ε, πλαισιώσουμε όλες τις απαραίτητες λύσεις. Γιατί πέρα από την 21η διάσκεψη των μερών στο Παρίσι, την COP21, θα πρέπει να κάνουμε το παν έτσι ώστε η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι ιδιώτες, οι επενδυτές να ε, συμβάλλουν, να επιτρέψουν με τη δράση τους την ανάπτυξη τέτοιου είδους μεταφορών και κυρίως αστικών μεταφορών. Και τέλος, ε, ο οικονομικός φάκελος. Το οικονομικό θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα είναι άλλωστε και ο ακρογωνίος λίθος της Συμφωνίας των Παρισίων. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε το παν και σε αυτό το πεδίο, ώστε για τους λόγους που παρουσιάζω στην έκθεσή μου, ώστε να έχουμε ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο που θα δοθεί στις χώρες ε, τις αναπτυσσόμενες για να μπορέσουν να αναπτύξουν τρόπους μεταφοράς πολύ πιο αηφόρους. Είναι οι αναδυόμενες οικονομίες, οι αναδυόμενες ε, χώρες που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας, έχουν ανάγκη το πράσινο ε, ταμείο. Θέλουμε να εγκριθούν 100 δις δολάρια ε, για αυτές τις ε, χώρες που βρίσκονται σε λεπτή, σε ευαίσθητη κατάσταση για να καταπολεμήσουν την αλλαγή του κλίματος. Και ο κλάδος των μεταφορών και σε αυτό το τομέα και σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές έχει τεράστια σημασία. Η 21η διάσκεψη των μερών θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για ένα άλλαγμα μοντέλου. Το ξέρουμε αυτό και σε επίπεδο κυκλικής οικονομίας και σε επίπεδο οικονομίας που συνδέεται με τις μεταφορές Θέλουμε μια νέα οικονομία σε ε, σχέση με τις μεταφορές και είναι ευκαιρία η 21η διάσκεψη των μερών να αποτελέσει σημείο καμπής για να είμαστε σε θέση να πούμε στις νέες γενιές, στο, στο μέλλον, στους νέους ανθρώπους ότι όχι μόνο το Δεκέμβρη στο Παρίσι, το, στα τέλη του 2015 ε, καταπολεμήσαμε την κλιματική αλλαγή και καταφέραμε να μην αυξηθεί η θερμοκρασία παραπάνω από δύο βαθμούς ε, παγκοσμίω, αλλά να είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτή η αλλαγή ε, μοντέλου οικονομικού μοντέλου ε, έγινε χάρη στην 21η διάσκεψη των μερών για μια οικονομία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Και περνάμε λοιπόν στο πρώτο πάνελ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον Κλάου Ζάιπ από το Ινστιτούτο Βούπερταλ, τον Hans Μπρένιξ ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τον ε, κ. Λίμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Γενική Διεύθυνση MOVE. Ε, έχετε λοιπόν 10 λεπτά ο καθένα το λόγο. Ξεκινάμε με τον κύριο Κλάους Ζάιτ. My name is... You just heard my name, Klaus from the Wuppertal Institute. Klaus λοιπόν, από το Ινστιτούτο του Wuppertal, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ερεύνης βιωσιμότητας στη Γερμανία, εξετάζουμε διαρκώς τις διαδικασίες της κλιματικής αλλαγής, τις περιβαλλοντικές αλλαγές, σχετικά με αυτήν την έννοια των πλανητικών ορίων. Και στην παρουσίασή μου θα σας εξηγήσω το ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις ερχόμενες δεκαετίες. Αυτό που τώρα γνωρίζουμε είναι ότι για να προσεγγίσουμε το στόχο των δύο βαθμών Κελσίου μας χρειάζεται μια μεγάλη κλίμακα ε, κοινωνική και τεχνολογική μετατροπή. Δεν θα είναι απλώς και μόνο η τεχνολογική πρόοδος. Θα χρειαστεί μια βαθύτατη αλλαγή και το τομή σε όλο το κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό σύστημα. μπορούμε να δούμε καταρχάς κάποιες ε, τάσεις, κάποιες απεικονίσεις τάσεων και κάποιες προβολές. Και ο κύριος ε, Μπρούνιγκς θα συνεχίσει με περισσότερα στοιχεία του ευρωπαϊκού επίπεδου στην επόμενη παρουσίαση, αλλά σε αυτό το γράφημα βλέπουμε μια έντονη αύξηση από 2,8 γιγατόνους από το 1970 μέχρι το 2010 που έχουμε στοιχεία ως τους 6,77 γιγατόνους. Δηλαδή μια τεράστια αύξηση λόγω της παγκοσμιοποίησης, λόγω διευρυγμένης οικονομικής ανάπτυξης και από ό,τι φαίνεται σε σχέση με αυτά που κάνουμε προς το παρόν, όπως και με την πράσινη ανάπτυξη, είναι ότι κινούμαστε. Έχουμε καινοτομία, έχουμε νέα πρότυπα επιχειρηματικότητες, έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα και αυτό οδηγεί σε νέες τάσεις και σε νέα ζήτηση. Αυτά είναι κάποια μεγέθη του τομέα των μεταφορών από το 2010 σύμφωνα με την έκθεση IPCC 27% ήταν η συμμετοχή και οι προβολές μας λένε ότι από το 6,7 θα πάμε στους 12 γιγατόνους ισοδύναμου διοξιδίου μέχρι το 2050. Και αυτό κυρίως ε, λόγω των διαφόρων δραστηριότητών μας, δραστηριοτήτων μας, με συγχωρείτε. Και θα πρέπει να, να διοργανωθούμε. Γιατί έχουμε όλο και περισσότερα οχήματα σε παγκόσμια κλίμακα, το οποίο εξωθεί κυρίως τα πράγματα. Τουλάχιστον ως προς τις εκπομπές διοξιδίου, γιατί εκτός από αυτές έχουμε και τις έμεσε εκπομπές, λέει ο μιλητή, οι οποίες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες συνολικά. Η εκτίμηση κόστου προέρχεται από την Παγκοσμία Τράπεζα και όταν σχεδιάζουμε οποιαδήποτε μετατροπή του συστήματος μεταφορών εξετάζουμε το κόστος, την οικονομική πτυχή. Ε, τουλάχιστον για το οδικό δίκτυο η, τράπεζα, η Παγκοσμία Τράπεζα εκτιμά ότι θα χρειαστούμε 70 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια ανά τόνο και ανά χιλιόμετρο και ανά έτος για να αναπροσαρμόσουμε το σύνολο των υποδομών. Αυτά είναι, αυτές είναι κάποιες εκτιμήσεις ειδικών, αλλά μας δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις και στο Παρίσι θα αφορούν και ποια σημαντικά τμήματα προϋπολογισμού θα χρειαστούμε για να κάνουμε, να πραγματοποιήσουμε μόνο τις τεχνικές αλλαγές. Και αυτό σας λέω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην τεχνολογική πρόοδο. Υπάρχει στην επόμενη διαφάνεια αν θέλετε ευχαριστώ Hans η διαφάνεια αυτή δείχνει τα κοινά μας θέματα συζήτησης ότι χρειάζεται μία αλλαγή παραδείγματος, μία αλλαγή προτύπου Και ο περιορισμός κινητικότητας βεβαίως δεν είναι επιλογή. Αργότερα θα σας δείξω και μια άλλη απεικόνηση για το πώς θα μπορούσαμε να το ξανασκεφτούμε αυτό το περί περιορισμού της κινητικότητας στις μεταφορές. Εν πάση περιπτώσει εδώ μιλούμε για τις μεταφορές εμπορευμάτων και με την ψηφιοποίηση και την απελευθέρωση της αγοράς και τις επενδύσεις ε, στις ε, υποδομές μεσοπρόθεσμα προτιμάται ακόμα το οδικό δίκτυο των μεταφορών. Γιατί με την ψηφιακή τεχνολογία είναι πιο ευέλικτο από τις, τους σιδηροδρόμους και τις ε, θαλάσσιες μεταφορές αλλά και εκεί κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις προκειμένου να καταφέρουμε να αλλάξουμε το σύστημα. Τώρα θέματα που πρέπει να τεθούν και στο Ινστιτούτο αρκετοί από εμά εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα θέματα κάποιοι έχουν εστιαστεί στα των αερομεταφορών, άλλοι στα οδικά, άλλοι στα σιδηροδρομικά και ούτω καθεξής. Και συμφωνώ με τον κύριο Σέλεν Χούμπα ότι χρειαζόμαστε ένα περιορισμό ορίου ταχύτητας της κλιματικής αναθέρμανσης και είναι πρόβλημα κατά την άποψή μας ότι αυτός ο στόχος των δύο βαθμών Κελσίου δεν συμπεριελήφθη στο σχέδιο EDP για το Παρίσι για τον τομέα των μεταφορών. Επίσης, θεωρούμε προβληματικό ότι θα πρέπει να βλέπουμε συνολικότερα το θέμα των εκπομπών και τις εκπομπές για παράδειγμα οξυδίων του αζότου γιατί όλες αυτές οι διαδράσεις ενός περίπλοκου συστήματος εκπομπών προκαλούν τη θέρμανση του πλανήτη και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε κάπως λεπτομερέστερα. Επομένως η τεχνολογική αλλαγή είναι αρκετή επαρκεί στο να αντισταθμίσει την όλο και ευξανόμενη ζήτηση μεγαλύτερης κινητικότητας που έχουμε στη σύγχρονη κοινωνία μας. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα στη Γερμανία, για παράδειγμα μέσω των ηλεκτρονικών οχημάτων και μεγάλων επιχορηγήσεων σε αντίστοιχα έργα ηλεκτρικής κινητικότητας. Δεν εξαρτάται λοιπόν πάντα από την τεχνολογία αλλά και από τις κοινωνικές διαδικασίες και τάσεις. Όταν χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό όχημα πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά σε κάποιες καθημερινές του ασχολίες και επομένως να δούμε και τον αντίκτυπο τον κοινωνικό υπό αυτήν την έννοια. Και τελικώς μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς να περιορίσουμε τη ζήτηση για περισσότερη κινητικότητα Δηλαδή ένα μελλοντικό σύστημα σε τι θα πρέπει να εστιαστεί στην απόσταση, στην οικονομία κλίμακος σε σχέση με τις μεταφορές και τον τρόπο που θα πρέπει να πραγματοποιούνται. Χρειαζόμαστε πέραν αυτών μια κοινωνική αλλαγή και μια καλύτερη διαχείριση για να μην πω μετατροπή ή μεταρρύθμιση της ζήτησης για την ε, κινητικότητα. Δεν είναι θέμα μόνο τεχνολογία. Σα ευχαριστώ και που τηρήσατε και το χρονικό όριο και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Hans Brönix από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τι τελευταίε εξελίξεις και τα τελευταία πορίσματα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματο, τι εκπομπές διευθυντή του άνθρακα και σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ. Θα εστιαστώ σε τρεις εργασίε τη Υπηρεσία. Καταρχάς, η έκθεση τάσεων και προβλέψεων που δημοσιεύτηκε την περασμένο μήνα που παρακολουθεί τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερον, η έκθεση για τις μεταφορές και για το περιβάλλον που θα δημοσιευτεί πριν από το νέο έτος και τα στοιχεία, τα αναφερόμενα των ε, αυτοκινητών παραγωγών που περιλαμβάνονται, αλλά η υπηρεσία μας κοιτάει και πιο πέρα στο μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι εργαζόμαστε επί μίας έκθεσης για μίας μεγάλης κλίμακας εξέλιξης και προόδου του ηλεκτρονικού, της ηλεκτρονικής οδήγησης και της, ε, των επιπτώσεων που θα έχει στις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Κοιτώντας τους ε, στόχους στην Ευρώπη, ο συνολικός στόχος σε ό,τι αφορά τις τα του θερμοκηπίου για το 2030 είναι ότι θα είναι 8% πιο πολύ από ό,τι στη δεκαετία του 90. Αυτό μπορεί να θεωρήσετε ότι αποτελεί αύξηση, αλλά είναι, κάτω, είναι παραπάνω από 20% πιο χαμηλό από το ποσοστό που ήταν στις ε, εποχές ε, κορυφαίας εκπομπής. Για όσους ε, κοιτάτε λοιπόν το γράφημα, αυτό τι σημαίνει ότι το γράφημα σε ό,τι αφορά την καμπύλη απαλλαγής από τον άνθρακα θα πρέπει να επιταχυνθεί μέχρι το 2050. Αυτό ασφαλώς αποτελεί σημαντικό, σημαντική πρόκληση. Σε ό,τι αφορά τώρα το στόχο για την αυσιπλοεία, μιλάμε για μείωση 40% σε σχέση με το 2005 μέχρι το 2050 δηλαδή. Και αυτό αποτελεί σοβαρή βελτίωση γιατί από την δεκαετία του 90 έχουμε παρατηρήσει αύξηση 30 σχεδόν 100 στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό σε ό,τι αφορά τους στόχους. Τώρα, αυτό που είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε είναι η, την μεταφορά και την ε, κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου και σε σχέση με τους άλλους τομείς. Βλέπετε λοιπόν στην κορυφαία καμπύλη τον τομέα των μεταφορών. Είναι ο μοναδικός τομέας στην Ευρώπη που από τη δεκαετία του 90 έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είμαστε συν 20% σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Και η αεροπορία έχει διπλασιαστεί από τη δεκαετία του 90 και στην αυθυπλογή έχουμε συν 40% όπως σας είπα. Όπως βλέπετε από το 2007 και μετά υπάρχει μια πτωτική τάση. Το 2007 ήταν το έτος με τις υψηλότερες ε, ε, τιμές. Αυτό και λόγω νομοθεσία και λόγω συμπεριφοράς ε, των καταναλωτών, των νεαρών, αν θέλετε, πολιτών και κατά τρίτον και η οικονομική κρίση επέξε το τη για το 2014. Εκτιμούμε ότι θα σταματήσει αυτή η πτωτική τάση και αναμένουμε ελαφρία άνοδο των τιμών ε, για το 2014 και να μην συνεχίσει αυτή η πτωτική τάση μέχρι το 2030 ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Και αυτό ασφαλώ δεν συνάδει με του στόχου που έχουμε θέσει και του οποίου συζητήσαμε πριν από ένα λεπτό. Αν τα συγκρίνουμε λοιπόν όλα αυτά και με του άλλου τομεί, βλέπουμε ότι και πάλι επαναρχόμαστε σε μια οικονομία, σε μια κοινωνία απορριμμάτων. Στι μεταφορέ, λοιπόν αυξάνονται ακόμα οι εκπομπέ. Τα επιβατηγά πάνω από 40%, 43% συγκεκριμένα τα φορτηγά και τα λεωφορεία 13%, ε, τα μικρά φορτηγά 8,3%, τα επιβατικά από ό,τι ξέρουμε ρυθμίζονται, υπό σε ρύθμιση από το 2009 και τα μικρά ε, βάν από το 2011, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ε, νομοθεσία για τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς από εσά είναι ότι η διεθνής αεροπορία είναι στο 12% σε ποσοστό 12% των εκπομπών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διεθνή αεροπορία είναι στο 12% περίπου. Αυτό λοιπόν ε, είναι κάτι το οποίο θα μας πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον, όπως ξέρετε. Ε, τα πιο πολλά από αυτά εμπίπτουν σε τομείς που δεν είναι στο ETS. Κοιτώντας τώρα τις ε, νομοθετούμενες εκπομπές από νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη μειώνονται. Αλλά αυτά είναι σε συνθήκες ε, εργαστηρίου. Το περασμένο έτος λοιπόν αυτό φαντάζομαι ε, δεν σας θύμισε τίποτα, αλλά τώρα νομίζω κάτι σαφές σημαίνει αυτό πλέον. Και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση καυσίμων υπολογίζουμε 20-30% περισσότερο. Το βλέπετε κι εσείς όταν οδηγάτε τα αυτοκίνητά σας. Σε ό,τι αφορά τον NOx τώρα, εκτιμάτε... Βλέπουμε λοιπόν ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης. Τα στοιχεία τα οποία σας παρουσιάζω εδώ βασίζονται στα νέα μοντέλα του κάθε έτους και τα παρακολουθούμε μιας και όλοι οι παραγωγοί αυτοκινήτων αν μας παρέχουν τα στοιχεία αυτά. Το 2014, 53% των αυτοκινήτων που πουλούνταν στην Ευρώπη ήταν δίζελ, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι αν ξεκινήσουμε το 2000, η πάνω γραμμή είναι τα πετρελαιοκίνητα και τα... η δεύτερη γραμμή είναι τα αυτοκίνητα diesel. Η διαφορά λοιπόν που υπήρχε και ήταν πολύ έντονη στην αρχή, με την πάροδο του χρόνου έχει μειωθεί σημαντική αυτή η τάση γιατί γίνονται διάφορες εικασίες και διάφοροι μίσοι επικρατούν σε ό,τι αφορά τους δύο κινητήρες, τα δύο είδη κινητήρων. Κοιτώντα τώρα τι γίνεται με την πολιτική και τις προοπτικές. Ασφαλώς σήμερα ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε στόχους για το 2020-2030, ενώ εν γέννη η γενικότερη τάση καταδεικνύει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μπροστά από τους στόχους, πάνω από τους στόχους. Άρα πετυχαίνουμε τους στόχους πολύ πιο πριν από τις προθεσμίες, έως τώρα. Κοιτώντα τι γίνεται και τι προβλέπεται για το μέλλον, το 2030 μιλάμε για 95%, 95 διεξίδιο του άνθρακα ένα χιλιόμετρο, ε, ε, εκτιμούμε ότι αυτό τον στόχο θα το πετύχουμε πιο γρήγορα. Αλλά αν κάνουμε ένα άλμα μέχρι το 2050, εδώ μιλάμε για 60% μείωση στον τομέα των ε, αερίων του θερμοκηπίου, όπως αναφέρθηκε στη Λευκή Βίβλο. Εδώ λοιπόν αντιμετωπίζουμε με μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ξέρουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να το πετύχουμε με προσαρμογή των κινητήρων καύσης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιος θα φτιάξει λοιπόν το αυτοκίνητο του μέλλοντος, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι Google, οι Amazon, αυτόν του κόσμου. Αυτοί θα κάνουν την επανάσταση του μέλλοντος όπως συνηθίζουν και κατά δεύτερον υπάρχει και το επιχειρηματικό μοντέλο. Όταν αγοράζουμε αυτοκίνητο ξέρουμε από το GPS και από άλλες ε, συσκευές ότι ένα αυτοκίνητο το χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης 8% του χρόνου και 2% του χρόνου ψάχνει πάρκινγκ. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο θέλουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο του μείον 60% μέχρι το 2050. Υπάρχουν Ε, μάρκες όπως η BMW, οι οποίες βγάζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 400, ε, 450 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κοπενχάγη σήμερα, μέσω ενός συστήματος ε, κοινή χρήσης αυτοκίνητων. Αυτό είναι καλό και για τις επιχειρήσεις, γιατί και πολλούν και πολλά αυτοκίνητα και πλασάρουν μια κάποια εικόνα που προσελκύει τους νέους αν και αυτό ασφαλώ ε, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενδεχομένω να φτιάχνετε. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο σύστημα κινητικότητα και μετακίνηση θα επικρατήσει στο μέλλον και φυσικά το αυτοκίνητο θα δραματίσει σημαντικό ρόλο. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε τέτοιου είδου συστήματα για το μέλλον, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή η Ευρώπη θα προετοιμαστεί για μια τέτοιου είδου ε, ε, αλλαγή των μεταφορών που θα χρησιμοποιούν φυσικά και το αυτοκίνητο, αλλά σε συνεργασία, σε συνδυασμό και με άλλους τρόπους μεταφορών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πόλεις και τους, τον νέο κόσμο. Κατά πόσον λοιπόν θα προετοιμαστεί η Ευρώπη για αυτού του είδους την ανταγωνιστικότητα ή κατά πόσον θα μείνει κολλημένη σε μια παλιά τεχνολογία η οποία κάθε μέρα νομίζω αποδεικνύει τα όρια της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, όλα και πρόεδρος, κύριε Μπράνινγκς, Ο Ρόλφ Ντίμα από την Γενική Διεύθυνση MOVE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Hello, Mr. Chairman. Γεια σας, ε, κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ, τον Πίτερ Βίμαντ. Λέγομαι ε, Βις. Νομίζω ότι είχατε ήδη αυτό το νέο, δεν ξέρω αν ε, δεν σας το διαβίβασα. Ο πρόεδρος διακόπτει και λέει «Με συγχωρείτε που έκανα λάθος το όνομά σας και εσείς βεβαίως είστε πρόσδεκτος». Να σας εξηγήσω ποιος σας μιλάει. Έχω εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 χρόνια, κυρίως για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ήμουν επικεφαλής του προσωπικού και πολιτικού γραφείου της Κόνη Χίντεκαρτ, της Επιτρόπους, κατά την προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Και αυτή τη στιγμή εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση MOVE. Είμαι ο μόνος που εργάζομαι αποκλειστικά και μόνο για το decarbonization, μια οικονομία που θα εξαρτάται όλο και λιγότερο από τον άνθρακα. Και δουλεύω εγκάρσια σε σχέση με και σε συνεργασία με όλες τις γενικές διευθύνσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα ήθελα να σας πω το πλαίσιο Τη συνάντηση των Παρισίων. Εγώ ήμουν διαπραγματευτή τη διασκέψη των μερών όταν αυτέ είχαν μονοψήφιο αριθμό και τώρα έχουμε φτάσει στην 21η. Περίπου 150 χώρε έχουν ε, υιοθετήσει δεσμεύσεις πολιτικές, όρκους πολιτικούς να σας το πω έτσι και ο επίσημος όρος είναι εκ προθέσεως εθνικώς αποφασισμένες συνεισφορές, τα INDCs δηλαδή, Περί τίνος πρόκειται. Είναι δέσμευση πολιτική που υιοθετεί ε, χώρα, οποιαδήποτε χώρα, να υιοθετήσει πολιτικές που θα είναι υπέρ του μετριασμού της ε, κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα ήδη. Πριν φτάσουμε στο Παρίσι, έχουμε ήδη ένα πολύ ευρύ φάσμα δεσμεύσεων πολιτικών από χώρες κάθε μία ξεχωριστά. Πολύ περισσότερες πολιτικές δεσμεύσεις από αυτές που είχαν υπάρξει την εποχή του πρωτόκολλου του Κιώτο, όπου οι εκπομπές που καλύπτονταν ήταν μόνο το 12% επί του συνόλου. Έχουμε φτάσει από το 12% στο πρωτόκολλο του Κιώτο στο 90% σήμερα, ακόμα και πριν το Παρίσι, στις παραμονές του. Και αυτό ήδη μεταφράζεται σε πρόοδο. Η Ευρώπη έχει δεσμευθεί να μειώσει κατά 40% ε, μέχρι το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 την εξάρτησή της από τον άνθρακα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσει ε, πολιτικές συγκεκριμένες, ενώ θα χρειαστούν και νέες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αξιοποιηθεί η πλειάδα εργαλείων και μηχανισμών, όπως είναι τα πρότυπα διοξιδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα, όπως είναι το σύστημα εμπορίας ρήπων, εκπομπών, όπως είναι τα ε, αέρια τα φθορίζοντα με βάση το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που χρησιμοποιούνται σε κινητά ε, συστήματα κλιματισμού διάφορα τέτοια πρότυπα, συστήματα και εργαλεία έχουν υιοθετηθεί που έχουν διαφορετικό αντίκτυπο το καθένα σε διαφορετικούς υποτομεί του κλάδου των μεταφορών. Πρόκειται όμως για ένα άθροισμα πολιτικών και θα πρέπει αυτές και να επεκταθούν και να διευρυθούν και να ενισχυθούν στο μέλλον. Οι οδικές μεταφορές κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν και το βασικό, ο βασικός τρόπος μεταφοράς και στο μέλλον στην Ευρώπη. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μειώσει ή να να εξαλείψει την εξάρτηση της αυτοκινητοβιομηχανίας από τον άνθρακα, ε, προωθώντας εναλλακτικά καύσιμα ή την ηλεκτρική ενέργεια και, την, και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφοράς των συγκοινωνιών και αυξάνοντας τα πρότυπα, τα στάνταρ διοξιδίου του άνθρακα για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Θέλουμε να, ε, μετα, να κάνουμε μια μετατροπή, μια μεταστροφή προς λιγότερο ρηπογόνους τρόπους μεταφοράς όπως είναι οι, οδη, οι ε, μεταφορές και οι μεταφορές μέσω ε, εσωτερικών υδάτινων οδών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη σωστή υποδομή και αυτά να τα στηρίξουμε ε, οικονομικά. Αυτό απαιτεί συμπληρωματικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. Την ενθάρρυνση καθαρών δημόσιων μεταφορών και την ενθάρρυνση της ποδηλασίας βεβαίως. Πρέπει να επανεφεύρουμε την κινητικότητα. Πρέπει να έχουμε καινοτομία και ευφυείς τεχνολογίες και έτσι θα στηρίξουμε έξυπνα και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς και θα διαχειριστούμε καλύτερα τη ζήτηση για μεταφορές και ανθρώπων και αγαθών, ακόμα και ε, σε αστικές περιοχές. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα ανελιπώς κάθε χρόνο από το 2002 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια εκστρατεία η οποία χρησιμοποιεί το λογότυπο της διάσκεψης των μερών 21 και που θα προωθηθεί στο πλαίσιο ε, της Συνόδου των Παρισιών. Όμως, φέτος 1869 πόλεις ε, υιοθέτησαν και προσχώρησαν στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό στο Παρίσι είναι ότι η Σύνοδος των Παρισίων δείχνει ξεκάθαρα ποια κατεύθυνση πλέον να ακολουθούν οι ηθήνοντες πολιτικής, οι βιομηχανίες, που θα πρέπει να επενδύσει κανείς και αν μου επιτρέπετε ένα θέμα μεταφορά να θέσω που έχει τεθεί επιτάπητο στη διαπραγμάτευση στο Παρίσι είναι το εξή. Το διαπραγματευτικό κείμενο, το κείμενο υποδιαπραγμάτευση, έτσι όπω έχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αναφέρθει στην ανάγκη για το Διεθνή Οργανισμό πολιτική αεροπορία και για το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοεία και Ναυτιλίας να συμφωνήσουν για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τι διεθνεί μεταφορέ, γιατί αυτό ο κλάδος είναι που ευθύνεται όλο και περισσότερο για αυτό το φαινόμενο. Αυτό είναι ένας από τους στόχους μας. Και θέλουμε οι δεσμεύσει πολιτικής που υιοθετούν οι χώρες, οι εθνικές συνεισφορές, το TINDCs, να μην σταματήσουν στο Παρίσι, αλλά να υπάρχουν κανόνες επαρκούς λογοδοσίας και διαφάνειας, έτσι ώστε κάθε χώρα να εφαρμόζει μια πολιτική και να μπορεί ο καθένας να επιβεβαιώνει ότι πράγματι δουλεύει η πολιτική της. Δεν χρειαζόμαστε ε, τόσο πολλά λόγια όσο πράξεις. Άλλωστε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίως είναι ε, σταθερά προσιλωμένοι ε, στους κανόνες λογοδοσίας και διαφάνειας και θέλουμε αυτά να χαρακτηρίσουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι. Αυτά κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ω τώρα λοιπόν έχουν ζητήσει το λόγο τρία άτομα Κριστίνα Ριμπουνταλόν, Βέρεν Κούν και Μάρκο Πίπερ. Ladies first. Merci, merci, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωτοβουλία αυτή αυτής εδώ της συνάντησης είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Το γνωρίζαμε και το επιβεβαιώσατε. Ο τομέας των μεταφορών προκαλεί τη μεγαλύτερη ρήπανση. Αλλά αυτά που προτείνεται θα χρησιμεύσουν για να υλοποιήσουμε τη φιλοδοξία μας, να μετατρέψουμε τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε και μεταφέρουμε σήμερα και όλα τα συμπληρωματικά που μπορούμε να κάνουμε εν είδη κυρώσεων, αλλά επιπλέον ως κινητήριος μοχλός ώστε να αλλάξουμε τα πράγματα στους βασικούς κλάδους βιομηχανίας όπως ο αυτοκινητιστικός. Δηλαδή να το δούμε σαν μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τα πράγματα γιατί όπως είδαμε στις παρουσιάσεις είχαμε και μια εχμή το 2007 αλλά μετά ακολούθησε μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα θετικό μήνυμα ενδεχομένως και για το στόχο που ανέφερε η Κομισιόν του 40% και πρέπει να τον επιτύχουμε πολύ συγκεκριμένα τι χρονοδιάγραμμα θα ακολουθήσουμε γιατί το είδαμε και το πρωί όλα τα προβλήματα αυτά στις μεταφορές απασχολούν όλους αλλά πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις απτές θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε όλα αυτά όχι ως τροχοπέδι για την οικονομία, αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε ακόμα περισσότερες καινοτομίες ε, μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να σκεφτούμε και να υλοποιήσουμε για να ηγηθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή της αλλαγής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βέρνης Κούν τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ζετ Μπράουνιξ και Φις. Η κατεύθυνση ήταν η ίδια και στις τρει ε, παρουσιάσει. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μειωθεί και να περιοριστούμε στους δύο βαθμούς. Η οικονομία η οποία ανθεί πάντα έχει κάτι να κάνει με τις μεταφορές. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αλλά βλέπουμε στις οδικές ε, μεταφορές Ποιο είναι ο μεγαλύτερος υπεύθυνο της εκπομπές. Η Επιτροπή Μεταφορών αυτό το έχει αποτυπώσει και έχει ασχοληθεί με την κατάσταση αυτή με διάφορες οδηγίες. 135 ε, γραμμαρία ανά εκπομπές, δηλαδή ακόμα και για μικρές ε, μεταφορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουν ε, ολόκληρα συστήματα, ολόκληρες γενιές τα επόμενα 10 χρόνια, προκειμένου να περιοριστούμε για να πετύχουμε ακριβώ αυτά τα 135 γραμμάρια, να περιοριστούμε στα 5 λίτρα κατανάλωση κλπ. Αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία μας από τον δρόμο στη θάλασσα, από τις ε, οδικές μεταφορές στις ε, θαλάσσιες μεταφορές και στις οδικές πλωτές μεταφορές ε, και στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η πιο ιδανική η κατανάλωση. Αλλά και αυτό λοιπόν θα πρέπει να λεφτεί υπόψη και αυτός ο όρος. Ύστερα έχουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές οι οποίες συχνά τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ε, ενέργεια και στις αεροπορικές μεταφορές έχουν επιτευχθεί προοδικές εξελίξεις, αλλά έχουμε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους ε, στη γη αυτή. Και το ΕΕΠ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 20%, αλλά η κατανάλωση ενέργεια μόνο κατά 5%. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά σωστά διευκρινίσατε ότι εξακολουθούμε να σπαταλάμε πάρα πολύ ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν ψάχνουμε θέση πάρκινγκ στην κίνηση. Ε, εργοστάσια καύση. Ε, όλα αυτά δεν μπορούν φυσικά να ακολουθήσουν την καμπύλη σε ό,τι αφορά την κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα όταν ε, κανείς για παράδειγμα ε, προχωράει στο αυτοκινητόδρομο, οδηγάει στον αυτοκινητόδρομο 200 χιλιόμετρα την ώρα, βλέπουμε πόσο μεγάλη κατανάλωση καυσίμων έχουμε. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν σημαντικά και καταστατικά ζητήματα. Ερωτώ λοιπόν, στοχευμένα, τι γίνεται με την τηλεματική σε ό,τι αφορά το δικό μας GPS, το Γαλιλαίο. Για είναι αποφυγή σημείων, ε, για παράδειγμα, μεγάλη κίνηση στον δρόμο Γιατί λίγο την κατανάλωση καυσίμων. Τι δυνατότητε έχουμε βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα, με νέα γενιά κινητήρε, όπω η υβριδική, αλλά και άλλοι για παράδειγμα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα για το εσωτερικό της πόλης, τι γίνεται με την έρευνα για την αποθήκευση ενέργειας, μπαταρίας λιθίου για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Ναι, με ρηκτό καύσιμο, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό και ευνοϊκό στην ε, κατανάλωσή του. Αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσει που έχω να κάνω σε ό,τι αφορά και τη μεσοπρόθεσμη διάσταση των οδικών, συνδρομικών και αεροπορικών μεταφορών. Σας ευχαριστώ και δυστυχώς επειδή ζήτησαν και άλλοι το λόγο θα πρέπει να σας περιορίσω στο δύο λεπτά τον καθένα. Είχαν δίκιο οι εκπρόσωποι του Μεκλεμού ο Μάρκο Πίπερ. Ναι, μετά από μένα. Μετά από μένα νομίζω ότι ξεκινάει το όριο του χρόνου. Αν σωστά κατάλαβα. Όχι, όχι. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και του ε, προσκεκλημένου για τι ιδέε που μα παρουσίασαν για την ε, εξοικονόμηση ενέργεια. Όλα αυτά είναι πολύ ωραίε ιδέε οι οποίε πραγματικά μα συναρπάζουν τεχνολογικά. Και προφανώ θα υπάρχουν και κίνητρα από την αγορά. Αυτό που με ενοχλεί και στις τρεις περιπτώσεις είναι οι αναλύσεις και όλα τα σενάρια. Ότι αν δεν συμβεί αυτό, θα συμβεί αυτό. Μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για μια δικτατορία παγκόσμια η οποία ε, καταλύει ουσιαστικά δημοκρατικές αρχές για να επικρατήσουν όλα αυτά που προβλέπονται. Και δεν θα ήθελα λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη λογική. Θα ήθελα να κάνω κάποιε ερωτήσει και να απευθύνω κάποιε ερωτήσει και προ του τρει ε, προσκεκλημένου. Καταρχά, ο στόχο των δύο βαθμών. πρέπει να σα πω ότι έκανα κλιματολογία στο Πανεπιστήμιο και τότε ε, έμαθα ότι μέσα από 15.000 χρόνια στη μία ανθρώπινη ζωή ε, η θερμοκρασία ενδεχομένω να και 4 4-5 βαθμού. Πώ θα αποφασίσουμε δηλαδή πολιτικά ότι θα πρέπει να περιοριστεί αυτή η αύξηση σε 2 βαθμού, δεν αμφισβητώ την επιρροή του ανθρώπου σε διαφορά του του άνθρακα. Μην με παρανοήσετε. Απλά λέω ότι μπορεί να προκληθούν πολύ πιο δραματικές αλλαγές. Ύστερα, για το ερώτημα του τι έχετε συγκεκριμένα υπόψη σας. Πολύ λυπάμαι, αλλά αυτές οι ερωτήσεις κινούνται προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Επιτρέπετε μου να τις κάνω. Είπατε ότι οι εκπομπές αυξήθηκαν. Αν το αναγάγουμε σε χιλιόμετρα ανά αυξήθηκε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, το diesel. Τι ακριβώς εννοείται. Τι είδους κινητήρες. Και τελευταία ερώτηση. Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για τον οικολογικό φόρο και το καθεξής. Αν τον είχαμε επενδύσει όλα αυτά για όχι σε κοινωνικές παροχές και συστήματα ασφάλειας, αλλά σε κοινοτομία, ε, έχετε υπόψη σας που θα βρισκόμαστε σήμερα αντί να επιβάρουμε διαρκώς νέα επιβάρυνση, νέες φορολογίες για να α, μπορούσαμε να απαλλάξουμε και λίγο από το βάρος του τον κλάδο αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, αλλά τα δύο λεπτά ισχύουν για όλους. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις που έθεσαν αλλά και τους ομιλητές. Νομίζω ότι μαζί με τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής πρέπει να μιλήσουμε και για τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, η οποία δολοφονεί περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες σήμερα από ό,τι συμβαίνει λόγω οδικών ατυχημάτων και ατυχημάτων στο τομέα των μεταφορών και της συγκοινωνίας γενικότερα. Είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαιτέρως και μετά την έλευση του σκανδάλου της Volkswagen πρέπει να δούμε όλο το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπασης το οποίο είναι τεράστιο. Οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δοκιμές στα αυτοκίνητα, οι οποίες γίνονται με συστηματικό τρόπο αντικείμενο χειραγώγησης, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει ότι σταματά ε, ε, προσωρινά τις εγκρίσεις και χρειάζονται αλλαγές για να έχουμε ένα παιχνίδι ίσης όρης. Και θα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη για να αλλαγές για να υπάρξει εμπιστοσύνη με, από τους ε, οδηγούς, τους ε, κατασκευαστές αλλά και τους επενδυτές. Προσωπικά να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι η Volkswagen τα έκανε αυτά μόνη της και ήταν η μόνη που τα έκανε αυτά. Νομίζω ότι και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να το έχουν κάνει και αν δεν κάνουμε κάτι ε, στην Ευρώπη θα χάσουμε από την Toyota και την Ιαπωνία. Θα ήθελα η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να ξυπνήσει, να ξυπνήσουν οι πολιτικοί και να κάνουν κάτι πριν είναι πολύ αργά και για τον κόσμο και για το, την αυτοκινητοβιομηχανία και για τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρενό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις διάφορες παρεμβάσεις. Δύο-τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω εν συντομία. Είναι σαφές ότι το τέλος των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα 300 δις στην Ευρώπη πρέπει πράγματι να διοχετευτεί ε, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώς θα γίνει αυτό, με ποιο μηχανισμό. Αυτό καταρχάς. Δεύτερον, βεβαίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ο καθένα έχει την ευθύνη για τη δική του χώρα. Μιλήσαμε για μια πολιτική ατζέντα ε, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, πώς μπορούν να αναλάβουν δράση. Τρίτον, οικονομικό πακέτο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει το project Lumière από τον κύριο Μπορλό για τον εξηλεκτρισμό της Αφρικής. Μπορεί αυτό να μπει στο οικονομικό πακέτο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Έχουν ε, Έχω βάλει και τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά αυτό το συναγερμό που ε, πρέπει να θέσουμε, γιατί δεν θέλουν να ε, υπερχειλήσουν και να βυθιστούν οι κάτω και να φτάσει η θάλασσα μου στο Βερολίνο. Θα ήθελα και εγώ να πω την άποψή μου και, και εγώ σα άφησα να μιλήσετε. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, κρούσουμε τον κόδωνα του συναγερμού. το δεύτερο. τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα κανονικό ε, όχημα, τα ευρετικά οχήματα. Αν ε, αληθεύουν αυτά που γνωρίζω, δεν ε, είναι πολύ καλύτερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα ήθελα να μας πείτε τι σχετικές τιμές. Τρίτο θέμα, Κοπεχάγη. Πριν από 25 χρόνια, αν σας έλεγα ότι στην Κοπεχάγη θα πηγαίνουν 53% ε, των ανθρώπων στη δουλειά τους κάθε μέρα μετά από την θα με λέγατε τρελό. Έγινε όμως. Έγινε σε αυτά τα χρόνια κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις πόλεις γιατί εκεί, από εκεί προκύπτουν 70% των βλάβερων εκπομπών. Έχουμε πολλά θετικά αποτελέσματα λοιπόν, πολλά θετικά παραδείγματα που προωθούν και την κινητικότητα και την προστασία του κλίματος και κάτι άλλο. Αν συνεχίσει να ισχύει αυτό. ο αθέμητος ανταγωνισμός. Αν υποστηρίζουμε τις ε, εκπομπές ε, ε, που βλάπτουν την, το περιβάλλον. Για παράδειγμα, στις αεροπορικές μεταφορές, στις δρομικές μεταφορές. Και στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσει όπου το 100% μιας ο ε, οδικός ε, επιβαρύνεται με δυο δύο, ενώ στου δρόμους είναι 0,9%. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον χρειάζεται σε θεμητός ανταγωνισμό για όλου. Οι ίδιοι, ίδιες συνθήκες για όλους. Να μην ε, επιβαρύνονται αυτοί που είναι φιλικοί προ το περιβάλλον και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Πίπερ που πήρε το λόγο για 7 δευτερόλεπτα παραπάνω. Έχετε το λόγο για 2 λεπτά ο καθένα για να απαντήσετε. I didn't know we... Δεν ήξερα ότι και για μα ισχύει ο κανόνας των δύο λεπτών. 17 ερωτήσεις πρέπει να απαντήσω. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ και συνεχίζω. Αν υπάρχει ένα το σχέδιο. Ναι, οι διάφορες πόλεις της Ευρώπης έχουν τελείως διαφορετική απόδοση στην υλοποίηση περιβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων. Έχουμε πολλά να μάθουμε στην Ευρώπη. Αν συγκρίνω την Κομπεχάγη με, την, με τις Βρυξέλλες θα μπορούσα να μιλάω για δύο ώρες, αλλά έχω δύο λεπτά. Έχουμε πολλή καινοτομία στην ε, βιώσιμη διοργάνωση της αλυσίδας του κλάδου των μεταφορών και εδώ έχουμε μεγάλη καινοτομία να επιδείξουμε και ηγούμεθα. Και όταν μιλάμε για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες με νέα μοντέλα αυτοκινήτων, νέες κινητήρες, νέες συστήματα ICT επιχειρηματικότητας υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Διότι η μετάβαση στα συστήματα κινητικότητας και στα οχήματα θα υποστηριχθεί και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου αυτή τη στιγμή η ποιότητα του αέρα στα αστικά κέντρα είναι τέτοιο πρόβλημα πολιτικό που η μετάβαση είναι αναπόφευκτη. Για το στόχο των 2 βαθμών Κελσίου δεν έρχεται από τους εθέρες αυτό. Επί τη βάση της IPCC και της επιστήμης τα τελευταία 2.000 χρόνια δεν έχουμε δει αλλαγές κλιματικές 4 ή 5 βαθμών Κελσίου αλλά υπήρξε μια σταθερή διαδρομή θερμοκρασιακή. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να δούμε τέτοιες κλιματικές μεταβολές με τέτοια ταχύτητα όπως παρατηρούμε σήμερα. Και αν δούμε την αποδοτικότητα την ενεργειακή απόδοση ενδεχομένως. Το διοξίδιο ανά χιλιόμετρο. Ναι, έχει κατέλθει στα αυτοκίνητα. Το ζήτημα είναι ότι κάνουμε περισσότερα χιλιόμετρα με περισσότερα και μεγαλύτερα οχήματα. Και η συνολική στόχη αποδοτικότητας δεν έχουν μεταφραστεί σε πίεση προς τον αυτοκινητικό κλάδο για τη μείωση του συνόλου των εκπομπών. Αν δείτε την ατμοσφαιρική ρήπανση. Πιστεύω όπως και είπε, είπε και η κυρία Κιούλερον ότι στην Ευρώπη έχουμε μια καλή ιδέα από πού προέρχεται η ρήπανση αυτή συμπεριλαμβανωμένη της κινητικότητας. Η εκτίμηση 400.000 πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη συνδέεται με θέματα ατμοσφαιρικής ρήπανσης όπως είχαμε πει και στην αναθεώρηση της δέσμης της ποιότητας ε, του αέρα. Για τις επιχορηγήσεις και τις επενδύσεις <clears throat> είναι σαφές ότι οι ενισχύσεις είτε άμεσες είτε έμεσες φορολογικές δηλαδή καθοδηγούν την αγορά και καθοδηγούν τις επιλογές των καταναλωτών που είναι ο βασικός παράγοντας εξήγησης της απομάκρυνσης από το ντίζελ του στόλου των αχημάτων στην Ευρώπη, αλλά σε πιο μακροσκοπικό επίπεδο θα έλεγα ότι οι ενισχύσεις προς το σύστημα που βασίζεται στον άνθρακα επί τη βάση της κινητικότητας είναι επιτάπητος και αυτό υποστηρίζεται από τον ΟΑΣΑ, από την Παγκόσμια Τράπεζα ε, πρόκειται για ένα ευρύ σώμα και πεδίο γνώσεως που έχει προκύψει για τις ροές ε, και την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ε, τεχνολογίας είναι σαφές, όπως είπε ο κύριο Κούν, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα διάθεσή μας για να έχουμε την καλύτερη απόδοση των πόρων, καλύτερη κατανομή, ευφυής διαχείριση της κυκλοφορίας. Έχουμε διάφορες τεχνολογίες και γνωρίζουμε ότι αυτές λειτουργούν, αλλά δεν εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα στις περισσότερες ευρωπαϊκές ε, περιοχές που έχουμε κυκλοφοριακό υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα υπάρξει υποστήριξη από τους πολίτες ενώ έχουμε αντίθετα παραδείγματα. Οι πολίτες είναι υπέρ των συστημάτων διαχείρισης της ροής που είναι καλύτερη και πιο ομαλή. Υπάρχει λοιπόν υποστήριξη από τους πολίτες. Θα μείνω εδώ προτού με κόψει ο Πρόεδρος στο δίλεπτο. να συνεχίσω εγώ λέμε ότι έχουμε δύο κατηγορίες έχουμε ε, ε, κατηγορίες ανθρώπων τους, του παρόντος και τους, του μέλλοντος ακούμε τα πορίσματα των θεωρητικών φυσικών που τα πορίσματά τους Τη υλοποιησιμότητας εμπαστός για το μέλλον τα τροφοδοτούν στα μοντέλα τους και μετά φτάνουν ε, στην υλοποίηση που πρέπει να γίνει ως προς το στόχο βαθμών Κελσίου ε, για μένα ως κοινωνιολόγος και πολιτικός επιστήμων σημαίνουν όλα αυτά ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν πολύ βραδύτερα γιατί τα κοινωνικά συστήματα και πολιτικά συστήματα κινούνται πολύ πιο αργά. Και προκύπτει η ερώτηση γιατί αυτές οι συναντήσεις υψηλού επίπεδου στο Παρίσι. Μήπως πράγματι εκεί αναλαμβάνουμε μια τεράστια, ένα τεράστιο πολιτικό εγχείρημα πηγαίνοντας κάθε λίγα χρόνια. Και τι έχει αλλάξει στην έρευνα βιωσιμότητες μεσοπρόθεσμα τα τελευταία χρόνια πάντοτε είχαμε συζητήσει επί της ενεργειακής απόδοσης. Αυτή είναι η μεσοπρόθεσμη στρατηγική. Αλλά αν δείτε του στόχους του Έλμαου που ήταν υψηλωτά του επίπεδου συνάντηση για την απομάκρυνση από τον άνθρακα την πλήρη μέχρι το 2100 και αυτό δεν είναι τόσο μακριά, είναι μια γενιά, 75 χρόνια. και μιλούμε για συνεχείς ε, μελέτες, ε, σενάρια, προβολές. Τι μπορώ να πω στο γιο μου που είναι δεκάχρονος, που θα ζει τότε. Πρόκειται λοιπόν για μια μετατροπή στις συζητήσεις μας. Πριν μιλήσουμε για βιωσιμότητα, η έρευνα αφορούσε στην ε, αποδοτικότητα και τώρα πλέον μιλούμε για την αναδιαχείριση του συνόλου του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος από το 2050 και μετά. Αυτή είναι έρευνα αλλαγής, απόλυτης αλλαγής, ακόμα και στο υψηλό πολιτικό επίπεδο. Ιδάλλως ε, μια συνάντηση του ΕΛΜΑΟ θα ήταν ψεύτικη. Σας ευχαριστώ και το συμμελητή ομιλητέ θα το ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, αξιότιμοι βουλευτέ, για τι ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις ε, νομοθετικές προτάσεις, για τις στρατηγικές ανακοινώσεις που προγραμματίζει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλώντας ε, για μια τεχνολογία σε ό,τι αφορά την, ε, τα οχήματα, τα καύσιμα των οχημάτων και τα συστήματα μεταφορών σε ό,τι αφορά την τηλεματική και σε ό,τι αφορά την πιο αποτελεσματική χρήση της, ε, των υποδομών. Το πρώτο ήμιση του επόμενου έτους θα έχουμε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την ε, χρήση λιγότερου ανθρακά στις μεταφορές. Και αργότερα, στο ίδιο έτος, θα γίνει αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας της φετινής για τα επιβατηγά οχήματα. Αυτό είναι το σχέδιο. Και θα υποβληθεί πρόταση για την παρακολούθηση και την εγκαταγραφή των εκπομπών από τα βαρέα οχήματα. Όπως γνωρίζετε, επίσης ε, συνεχίζονται οι εργασίες στους διεθνείς οργανισμούς, στον Διεθνή Οργανισμό Αεροπορίας για τις ε, εκπομπές της αεροπλοείας και μία οδηγία για τις εναλλακτικές αυτές μορφές μεταφορών που εγκρίθηκε πρόσφατα και περνάει από τα κράτη μέλη και θα περάσει στην Εθνική Νομοθεσία σύντομα. Προσπαθούμε λοιπόν να θέσουμε και τα πρότυπα για την αποτελεσματικότητα των οχημάτων και για θέματα διοξιδίου του άνθρακα σε συνάρτηση με την ενέργεια, προώθηση των καυσίμων, των αποδοτικών καυσίμων και της υποδομής που χρειάζονται και σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα των συσκευών τηλεματικής, γιατί αν δεν υπάρχει σύγκληση των τεχνολογιών, αν δεν προσπαθήσουμε να την προωθήσουμε, οι συσκευέ του αυτοκινήτου ενδεχομένω να μην μπορούν να επικοινωνούν με τι υπόλοιπε εκτό του αυτοκινήτου. Και προ την ε, κατεύθυνση αυτή εργάζεται λοιπόν η Γενική Διεύθυνση MOVE. Τέλο οι πραγματικές εκπομπές από την οδήγηση, ο έλεγχος των αυτοκινήτων. Αυτό, όπως ξέρετε, αποτελεί ένα νομοθέτημα που ψηφίστηκε σε επιτροπολογία τις τελευταίες ημέρες και τώρα λοιπόν θα περάσει από έλεγχο του Κοινοβουλίου. Κανονική διαδικασία λοιπόν υπό την επιτροπολογία και η βασική ιστορία είναι ότι ο κύκλος δοκιμής περιορίζεται και θα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω για την εξαρτησία των ελεγκτών, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Έχει ήδη ξεκινήσει. Τέλος, σε τοπικό επίπεδο αναφέρθηκαν οι καλέ πρακτικέ σε κάποιες χώρες όπως η ποντιλασία. Μπορεί να είδατε ότι στο σχετικό Συμβούλιο Μεταφορών τον Οκτώβριο αφιερώθηκε μία χρονοφυρίδα για την ποδηλασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να προωθήσει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, μεταξύ των πόλεων. Υπάρχουν ασφαλώ ε, τα οποία προκύπτουν, γιατί η ποδηλασία δεν χρειάζεται ασφαλώ απαραίτητα να ελέγχεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να ελέγχεται από το περιφερειακό επίπεδο. Αλλά προφανώ θέλουμε να διευκολύνουμε τέτοια προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ και ο κ. Μπράνινγκ ζήτησε να, να προσθέσει κάτι. Ναι, παρέλειψη να απαντήσω στην ερώτηση του, του Προέδρου για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα με εναλλακτικά καύσιμα και τις επιδόσεις του. Αυτό ίσχυε πριν από 15 χρόνια, δεν ισχύει όμως πια. Αντιθέτως, όλα αυτά τα αυτοκίνητα ε, βλέπουν τις βελτιώσεις τους να, επιδο... να... τις επιδόσεις τους να βελτιώνονται όλο και πιο γρήγορα και έχουμε πολύ μεγάλες ε, περικοπές και μειώσεις των, ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής, εσωτερικής καύσης. Άλλωστε θα πάμε προς το point source pollution και είναι πιο εύκολο να μειωθούν αυτές οι εκπομπές. Ακόμα και στη φάση μετάβασης δηλαδή, τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Όχι μόνο διότι έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα αυτοκίνητα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης ως προς τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις παρουσιάσεις και για την απαντήσεις. Στις 8 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών μας άκουσαν επί, τρει ώρε για την αστική κινητικότητα και το τι μπορεί να συμβαίνει η ποδηλασία και το ποδήλατο. Και ομόφωνα μετά από τρει ώρε αποφάσισαν να υπάρξει ειδικό χάρτη για το ποδήλατο. Και έτσι λοιπόν. Ε, συμφώνησαν ότι 50% των μεταφορών στις ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να γίνεται με ηλεκτρικά ποδήλατα. Φανταστείτε λοιπόν να πετύχουμε τέτοιες ε, επιτυχίες και γι' αυτό λοιπόν είμαι αισιόδοξος. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και ας περάσουμε στο επόμενο πάνελ. So, dürfte ich dann Sie bitten, Να σας παρακαλέσω λοιπόν να καθίσετε. Και περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα να καλωσορίσω. Πρόκειται για ένα πάνελ για τους ε, βασικούς τομείς μεταφορών. Τον Πέτρο Ντολίζιο θα ήθελα να καλωσορίσω από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση παραγωγών αυτοκινήτων, τον κ. Νέντμιν Χιούς, από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και τον κύριο Ντοτσιά, ε, τον εκτελεστικό του Clean Sky. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Πέτρε Ντολέζη. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Προσπάθη... Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να απαντήσω και σε ρωτήσεις στο τέλος. Καταρχάς να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία που θα πρέπει να συζητούνται πάντοτε όταν γίνεται λόγος για τις μεταφορές. Οι μεταφορές είναι απαραίτητες και για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και για τους ιδιώτες, είναι και για τη δημόσια υπηρεσία και για την ιδιωτική, μεταφέρουν αγαθά, παρέχουν υπηρεσίες, ε, είναι παράγοντας διευκόλυνσης της οικονομίας οι ιδιωτικές λύσεις επιτρέπουν κινητικότητα στο εργασιακό δυναμικό και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Και μάλιστα μας βοηθούν να προστατεύσουμε ε, ειδικέ κοινωνικές ομάδες έναντι της κοινωνικής συνοχής, συμπερίληψης, λέει ο μιλητής. Σε κάθε περίπτωση από το 2007 μέχρι σήμερα ακολουθούμε με συγκεκριμένη πορεία και θέλουμε αυτό να συνεχιστεί, γιατί πρέπει να επιτύχουμε κάποιους στόχους δύσκολους. δύσκολους. Και θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο ο ρυθμός είναι βραδύς ή κατά πόσο θα πρέπει να επιταχύνουμε. Οι μεταφορές λοιπόν έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην οικονομία και θα πρέπει να έχουμε παιχνίδι επίσης όρης μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Διαφορετική είναι η στόχευση και διαφορετικά, διαφορετικές οι απαιτήσει. Αν δούμε τις αλλαγές, πού ε, έχουν υποστεί οι διάφοροι τρόποι μεταφοράς, Βλέπετε ότι διευκολύνουμε, έχουμε τριπλασιάσει τις δυνατότητες μεταφοράς όχι μόνο με μέσω καραβιών αλλά και με, μέσω σιδηροδρομικής μεταφοράς. Μιλάω για τις εμπορευματικές μεταφορές. Ε, Συζητήθηκε και το σχετικό πακέτο στην Επιτροπή σας. Δεν ήταν εύκολη η συζήτηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση το να έχουμε ίσους κανόνες για όλους, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, η οικονομική προσβασιμότητα, να μπορεί κανείς να το πληρώσει. Πρέπει να έχουμε φανταστικές, φανταστικές λύσεις, αλλά να μπορεί ο κόσμος να τις χρησιμοποιήσει, ειδικά για τη μεταφορά των επιβατών. Κατά μέσο όρο το αυτοκίνητο στην Ευρώπη είναι 10 ετών και έχει τεχνολογία 10 ετών. Δεν σα ζητώ να εγκρίνετε επιδοτήσεις για να απολυθούν περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό θα βοηθήσει τη δουλειά μου βέβαια. Αλλά, αλλά αν βελτιωθεί ο στόλο, θα έχουμε πολύ μεγάλες βελτιώσεις και ε, στα περιβαλλοντικά θέματα. Αν διατηρήσουμε το στόχο 95 για άλλα 10 χρόνια, θα έχουμε ακόμα μείωση 30% των εκπομπών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν νέε λύσει και από πλευράς επιχειρήσεων και από πλευρά τεχνολογίας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέε λύσει σε υβριδικά αυτοκίνητα, σε λύσεις ε, ε, πολλαπλών τρόπων. Σίγουρα δεν γίνεται μόνο λόγος για την τεχνολογία. Ε, το θέμα είναι ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο που να μας βοηθά να εφαρμόσουμε ορισμένα μέτρα. Να μπορέσουμε δηλαδή να κατασκευάσουμε και να βάλουμε στους δρόμους σπουδαία αυτοκίνητα, αλλά να μην μένουν στον καράζ λόγω έλλειψης υποδομών. Ως προς το τομέα της ενέργειας, ναι, μπορούμε να τα βάλουμε να κυκλοφορήσουν στο δρόμο, αλλά αν για την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να κινηθεί το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται ορυκτό καύσιμο για να παραχθεί αυτή η ηλεκτρική ενέργεια, ε, τότε αυτό δεν ωφελεί και πολύ το περιβάλλον, έτσι δεν είναι. Μιλούμε λοιπόν για μια δέσμη μέτρων που θα πρέπει να υπάρξει. Και, για παράδειγμα, τα επιβατικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει γι' αυτά, ε, δίνεται έμφαση μόνο στη βελτίωση της τεχνολογίας. Ε, δεν αρκεί όμως αυτό, γιατί αναλόγως με τη δοκιμή βγάζει κάποιος 30 ή 40 διαφορετικά αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε λύσεις στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών για την οικολογική οδήγηση. Εμείς οδηγούμε τα μάξια, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό. Είναι μια συνολική προσέγγιση δηλαδή. Δεν είναι ε, μόνο το θέμα ο κινητήρας του αυτοκινήτου όπως και αν κινείται, με όποιο και αν καύσιμο και αν κινείται. Είναι μια συνολικότερη προσέγγιση που είναι απαραίτητη. Έχει ήδη υποθεί ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή του ITS Ξέρετε, την περασμένη εβδομάδα ήμουν στις κάτω χώρες και ξέρετε, είναι ωραία να είναι κανείς στα χωριά, αλλά υπάρχουν συγχρονισμένα φανάρια και αναγνωρίζει το φανάρι πότε έρχεται το όχημα και άρα το όχημα είναι υποχρεωμένο να σταματήσει. και τελικά με, το σωστό συγχρονισμό των φαναριών υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμων και ενέργεια γενικότερη. Ενώ αν γίνει αυτό στι Βρυξέλλε θα είναι πραγματικά κόλαση, να πρέπει κανεί να σταματήσει σε κάθε φανάρι. Χωρί συγχρονισμό δηλαδή δουλειά μας είναι να αξιολογούμε τις διάφορες λύσεις ε, κινητικότητας, συνεχώς προσπαθούμε να προσφέρουμε καινούριε λύσεις και αν συγκρίνω το στόλο των αυτοκινήτων με αυτόν που υπήρχε πριν από 10 χρόνια, οι αλλαγές είναι μεγάλες. Έχουμε υβριδικά αυτοκίνητα με ηλεκτρική μπαταρία αλλά και καύσιμο, έχουμε πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφέρουμε λύσεις με υγραέριο, πολλές και διαφορετικές λύσεις είμαστε σε θέση να προσφέρουμε. Όλοι ζούμε σε πόλεις και θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε λύσεις, αλλά πρέπει να πω και το εξής. Αναφέρθηκε ο ρόλος των πόλεων, ναι, όμως, αν έχουμε 200 διαφορετικές λύσεις στις πόλεις, θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Πρέπει οι πόλεις να υιοθετήσουν εναρμονισμένη προσέγγιση για να κάνουν οικονομία. Καλό είναι να εστιάζει κανείς στη βελτίωση του ντίζελ ή στην ηλεκτρική αγορά. Όμως είναι μικρή αγορά για μας. Και άρα υψηλό κόστος και άρα υψηλή τιμή για τον καταναλωτή. Τελικά δεν θα βοηθήσει αυτό κανέναν. Έχουμε εδώ την αρχή της επικουρικότητας και συμφωνώ. Εμείς όμως χρειαζόμαστε παγκόσμιες λύσεις γιατί είμαστε παγκόσμιοι κατασκευαστές και οι λύσεις σε αυτό το τομέα κατακαιρματίζονται ε, και σε επίπεδο νομαρχίας ή σε επίπεδο δήμου. Προσπαθούμε να προσφέρουμε λύσεις, ελπίζουμε ότι θα προσφέρουμε όλο και περισσότερες λύσεις και μπορώ να σας πω τώρα τι μπορούμε να προσφέρουμε σε σχέση με την 21η διάσκεψη των μερών στο Παρίσι. Έχουμε ήδη έτοιμο το κλιματικό και ενεργειακό παρεκέτο μας για το 2030 που θα αναθεωρήσουμε βέβαια μετά τη διάσκεψη των μερών αλλά ήδη υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο, πολύ σταθερό που μας δείχνει προς τα που πρέπει να πάμε και θεωρούμε ότι είναι πολύ φιλόδοξο συγκριτικά με τη ΣΥΠΑ ή με την Ιαπωνία. Ωστόσο, πρέπει να μην είναι μόνο φιλόδοξο, να είναι και εφικτό, να γίνεται να εφαρμοστεί και να τηρούν και οι υπόλοιποι τις δεσμεύσεις τους. Καλό είναι που εμείς θα φέρουμε αποτελέσματα εδώ στην Ευρώπη, όμως στην ιστοσελίδα των φίλων μας για τις μεταφορές και το περιβάλλον βλέπουμε την Ιφίλιο και βλέπουμε πώς κυκλοφορούν σε όλο τον πλανήτη οι εκπομπές των αερίων. Εάν λοιπόν εμείς φέρουμε αποτελέσματα εδώ στην Ευρώπη και δεν το κάνει η Κίνα, ε, θα μας έρθουν τα προβλήματα εδώ, σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Θα πρέπει η 21η διάσκεψη των Μερών να οδηγήσει σε δεσμευτικές λύσεις και δεν θα πρέπει η Ευρώπη να είναι για άλλη μια φορά αφελής. Θα πρέπει να έχει ίδιες φιλοδοξίες με τους λοιπούς, με τους άλλους. Γιατί για να σας μιλήσω ειλικρινέστατα, γιατί να θέλουμε εμείς να είμαστε εδώ αν άλλοι μας δίνουν πιο ευνοϊκές ε, συνθήκες και προϋποθέσεις. Εμείς που δραστηριοποιούμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως πρέπει να υπάρξει ένα σημείο ισορροπίας και ελπίζουμε μετά ότι μετά αν υπάρξει σημείο ισορροπίας αυτό μετά θα αποτελέσει μέρος και τη δικής μας πολιτική. Σας ευχαριστώ και σας γλίτωσα και ένα λεπτό. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ για το ένα λεπτό που μου γλιτώσατε. Ο Edmund Hughes από το Διεθνή Οργανισμό Ευσυπλοείας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, εκπροσωπώ εδώ τη γραμματεία του IMO και με χαρά να σας δώσω και τη δική μας άποψη σε αυτήν την ακρόαση που έχετε διοργανώσει σχετικά με τους κλιματικούς στόχους. Οι θαλάσσιες μεταφορές παραδίδουν περίπου το 90% του παγκόσμιου όγκου εμπορίου. Είναι βασικός κινητήριος μοχλός παγκόσμιου εμπορίου Ο ΕΜΟ και τα 171 μέλη του αναγνωρίζουν τις τεράστιες προκλήσεις κλιματικής αλλαγής όπως και τις κοινέ προσπάθειες που ε, πρέπει να καταβληθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Επί δεκαετίες έχουμε ηγηθεί αποφασιστικά στην προσπάθεια για ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο εντός του οποίου η ναυτιλία έχει γίνει πιο καθαρή και πιο ασφαλής εξακολουθώντας όμως να παρέχει έναν οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς αγαθών και επιβατών στα πλαίσια μιας βιώσιμης κοινωνίας. Μια ανάγκη μείωσης ε, των εκπομπών από την αυτιλία έχει αναγνωριστεί από τον ΑΕΜΟ. Είχαμε σταθερά βήματα το 1997 με την υιοθέτηση του πρωτοκόλου για την ε, αποτροπή των εκπομπών αερίων από τα σκάφη που διέπει το 95% των εκπομπών αυτή τη στιγμή και απαιτεί νέα σκάφη να αναφυγηθούν έως το 2035 και θα πρέπει να είναι ε, ε, πιο αποδοτικά περιβαλλοντικά κατά 30%. <coughs> Έχουμε υποχρεωτικές προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης και μέσω της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αυτές έχουμε πραγματικά ηγηθεί της προσπάθειας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Τώρα, η κατανόηση των τεχνικών και άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί σημαίνει ότι πολλές ναυτιλικές εταιρείες αυτή τη στιγμή αναγνωρίζουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν τα σκάφη τους, αλλά μειώνοντας και την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος τους. Αναπτύσσεται λοιπόν, αν θέλετε, μια κουλτούρα επιχειρηματικότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέχρι τη μείωση του ίχνου του άνθρακα που έχει κάθε ναυτιλιακή εταιρεία. Σύμφωνα με τα μεγέθη που έχουμε στην τελευταία μελέτη για τις εκπομπέ ε, αερίου θερμοκηπίου, η συνολική εισφορά τη παγκόσμιας ναυτιλία μειώθηκε από το 2,8 στο 2,2 παρά την σημαντική αύξηση στον όγκο και στην ε, δυνατότητα μεταφοράς ανασκάφος. Χρειάζεται βεβαίως περαιτέρω προσπάθεια καθότι οι εκπομπές ε, ε, διοξιδού του άνθρακα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά από 50 έως 250% μέχρι το 2050. από το Μάρτλαν 6 που υιοθετήθηκε το 2012 συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για μια ενιαία ε, υλοποίηση των διατάξεων αυτών για όλο το στόλο. Έχουμε και την Επιτροπή προστασία του Περιβάλλοντος του IMO, η οποία εξετάζει περαιτέρω ενεργή μέτρα μαζί με σύστημα ε, συλλογής δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου των σκαφών. Τώρα, τα τεχνικά, λειτουργικά ή δημοσιονομικά μέτρα λαμβάνονται στον ε, IMO και αναγνωρίζονται από το πρωτόκολλο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιώτο, όπου αναγνωρίζεται ο IMO ως οργανισμός ο αρμόδιος για την επιβολή των μέτρων αυτών από την διεθνή ναυτιλία. Και αξίζει να θυμίσει κανείς γιατί είναι έτσι. Εν μέρη, λόγω της προ... περιπλοκότητας της κατανομής εκπομπών από σκάφη σε χώρες. Η επιτυχή υλοποίηση μέχρι σήμερα σημαίνει ότι μόνο ο IMO έχετε διεθνή μέσα στη διάθεσή του προκειμένου να επιβάλλει τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς αυτοδιατάξεις. Η διεθνή ναυτιλία έχει ήδη ένα καθεστώς επιβολής του νόμου Port State Control λεγόμενο σχετικά με την επιβολή των διατάξεων του κρατουλημένα ώστε να μην έχουμε πιο ευνοϊκές διατάξεις κάποιων χωρών αντί άλλων. και θα μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές ανασκάφος ειδικά συγκρινόμενες με άλλα ε, είδη μεταφορών, με άλλους κλάδους μεταφορών, προκειμένου να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα θαλασσίων μεταφορών. Πέρυσι, 9,8 δισεκατομμύρια τόνοι ανταλλάχθηκαν μέσω εμπορίας ναυτιλίας και αυτό θα υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2030. Θα χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφορά των σκαφών, δηλαδή μεγαλύτερα σκάφη και περισσότερα σκάφη. Επομένω έχουν σημαντικό αντίκτυπο επί του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Ο IMO πάντως έχει υπηρετήσει πιστά την παγκόσμια κοινότητα, γιατί όπως δείχνει επιδόσεις μέχρι σήμερα, ο IMO μπορεί να καλύψει περίπλοκα προβλήματα, πολυδιάστατα και με πάρα πολλές διεθνείς ε, προεκτάσεις. Αλλά είναι οπωσδήποτε ο κατάλληλος φορέας για να συνεχίσει να καλύπτει το θέμα αυτό υπό την έννοια των εκπομπών της διεθνούς ναυτιλίας. Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή, Eric από το Clean Sky. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εύκολα φαντάζεται κανείς ότι το Clean Sky έχει να κάνει με την αεροπορία, την αεροναυπηγική και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Η ευθύνη της αεροπορίας σε ό,τι αφορά την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα ανθρώπινης προέλευσης είναι περίπου στο 3% σύμφωνα με τις διάφορες επιστημονικές παραδοχές για αυτού του είδους τις εκπομπές. Ωστόσο, η αεροπορία είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ραγδαία και ούτως ή άλλως το ποσοστό αυτό καθεαυτό απαιτεί δράση και είναι ένα ποσοστό που θα αυξηθεί σίγουρα στο μέλλον. Εδώ βλέπετε μια γραφική παράσταση από, από την ΑΤΑΓ, μια διεθνή οργάνωση, ομάδα δράσης για τις αερομεταφορές, Air Transport Action Group, και αυτό δείχνει την εξέλιξη των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα εάν δεν κάνουμε τίποτα από πλευράς τεχνολογικής, από πλευράς καυσίμων που χρησιμοποιούνται και το καθεξής. Αν αφήσουμε την κατάσταση ως έχει και αν αφήσουμε ε, την αεροπορία να αναπτυχθεί ε, σύμφωνα με τις προβλέψεις, δηλαδή κατά 4 και 5% ετησίως, έτσι θα έχουν οι εκπομπέ διοξίδιο του άνθρακα. Τώρα, βέβαια, είναι υποσυζήτηση οι προβλέψει αυτέ για το 2050 και κατά πόσο να είναι ακριβείς, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα είναι σταθερή η ανάπτυξη της αεροπορίας και των αερομεταφορών γενικότερα και η ανάπτυξη αυτή ελάχιστα έχει πληγεί από την κρίση του 2008 ή από οποιαδήποτε άλλη οικονομική μεταβλητή. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε, θα πρέπει κάτι να κάνουμε με διάφορους τρόπους και με διάφορα μέσα τεχνολογικά μεταξύ άλλων έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική τάση ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η ομάδα δράσης αυτή ε, ε, προσωπεί όλες τις αεροπορικές εταιρείες και όλους τους ε, κατασκευαστές μέσων αεροπορική μεταφοράς και θέλουμε να μειώσουμε τα, την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 κατά 20% και κατά 50% μέχρι το 2050. Είναι φιλόδοξη στόχη και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα για να τους επιτύχουμε. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε την Ευρώπη, την κατάσταση στην Ευρώπη και τους ε, στόχους τους που έχουν τεθεί από την ΑΚΑΡΕ, το Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Αεροναυπηγική Έρευνα. Είναι μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από τις δημόσιες αρχές, από ερευνητικούς οργανισμούς και από αεροπορικές εταιρείες εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε, δύο είναι οι ημερομηνίες σημαντικές, το 2020 και το 2050 και δύο διαφορετικοί είναι οι στόχοι, άλλος για το 20 και άλλος για το 50. Το 50 φαίνεται μια χρονιά μακρινή στον ορίζοντα. Όμως ε, η αεροπορία είναι ένας κλάδος όπου οι εξελίξεις είναι αργές. Δηλαδή δύο δεκαετίες χρειάζονται ε, για να ε, επινοηθεί μια τεχνολογία μέχρι να έρθει η στιγμή να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη πτήση. Εάν θέλουμε λοιπόν να δράσουμε για το 2050 θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή τη δράση από σήμερα. Εδώ έχουμε για το θόρυβο των εκπομπών. Έχουμε τις ακαθάριστες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά και μονοξίδιο του αζότου μόνο. Και βλέπετε αντιστοίχως τα νούμερα. 50% μείωση το 2020, 75% το 2050. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις εκπομπές του υπάρχοντος στόλου στο μισό. Αυτό σημαίνει ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες αεροπλάνων οι νέες τεχνολογίες θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε αυτή τη μείωση. Το Clean Sky, ο καθαρός ουρανός. Είναι ο επιχειρησιακός βραχίωνας, ο βασικός επιχειρησιακός βραχίωνας για να υλοποιήσουμε αυτή τη φιλοδοξία. Έχει υποθεί επανειλημμένος ότι η τεχνολογία δεν θα είναι αρκετή, συμφωνώ, αλλά χρειάζεται και αυτή για την επίτευξη των στόχων σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Ο καθαρός ουρανός είναι ένα τεχνολογικό πρόγραμμα, μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτείται κατά 5% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 5% από τον ιδιωτικό τομέα. Και είναι σημαντικό σε αυτόν τον, τον κλάδο της οικονομίας, αλλά όχι μόνο, τα πιο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που έχουν ποτέ ε, ξεκινήσει έχουν στόχους περιβαλλοντικούς και στόχους που έχουν να κάνουν με ανταγωνιστικότητα γιατί σαφέστατα στο μέλλον τα ανταγωνιστικά αεροσκάφη θα είναι αυτά που έχουν χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Στόχος είναι να έχουμε δείκτες πολύ σημαντικούς ώστε οι διάφορες τεχνολογίες να είναι μεταξύ τους συμβατές και έτσι να επιτύχουμε τις επιθυμητές μειώσεις πρώτα σε βάθος χρόνου 2020 και στη συνέχεια σε βάθος χρόνου 2050. 4 δις ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος Καθαρός Ουρανός, Clean Sky και θέλω να προσθέσω ότι και το υδρογόνο και τα ε, καύσιμα είναι πεδία στα οποία ε, δραστηριοποιείται το Clean Sky αλλά και το Biobase Industry ε, που ε, θα ασχοληθεί με την έρευνα στα βιοκαύσιμα. Ο καθαρός ουρανός έχει να κάνει με όλους τους επιστημονικούς τομείς, με όλα τα συστήματα, με όλα τα είδη εξοπλισμών των αεροσκαφών, ηλεκτρικά συστήματα, κινητήρια συστήματα, ε, δομές κατασκευαστικές του αεροσκάφους και μιλούμε για αεροσκάφη γενικής αεροπορίας, μιλούμε για μικρά αεροσκάφη από 20 επιβάτες, από 20 θέσεις μέχρι ε, τα Airbus, τα μεγάλα αεροσκάφη των μεγάλων ε, εταιριών. Στα δεξιά βλέπετε την τεχνολογική αξιολόγηση, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ερευνητικοί οργανισμοί ασχολούνται με την τεχνική αξιολόγηση και κάθε χρόνο αξιολογούμε κατά πόσο οι τυσέντες εξ αρχής ε, στόχοι, οι οποίοι απεικονίζονται λεπτομερώς ανά κατηγορία αεροσκάφους, ε, έχουν επιτευχθεί με τη τεχνολογία που έχει ε, εξελιχθεί ή όχι. Και τα καλά νέα είναι ότι οι στόχοι της πρώτης γενιάς του καθαρού ουρανού, ουρανού που εκτείνονται μέχρι του χρόνου θα έχουν επιτευχθεί μέχρι τότε και στη συνέχεια θα έχουμε τη δεύτερη γενιά στόχων στο ερευνητικό μας πρόγραμμα. Αυτές οι φωτογραφίες και εικόνες σας δείχνουν ε, ε, κάποιες δραστηριότητες ε, ε, ε εν πτήση είναι πολύ, πολύ δαπανηρές αυτές οι δραστηριότητες. Έχουμε ε, τους δείκτες, δυνατότητες που δείχνουμε εν πτήση ε, ζωντανά για τη μείωση των εκπομπών. Για τα αεροσκάφη μεσαίων αποστάσεων που καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος των αερίων μεταφορών ε, σήμερα, σίγουρα με αυτή τη τεχνολογία μπορούμε να πετύχουμε το στόχο του 40% ε, μείωση ε, το στόχο της μείωσης κατά 40% των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ο κλάδος συμβάλλει, η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατά 50% και έτσι καταλήγουμε σε νέα προϊόντα. Κάτι ωφέλιμο για την οικονομία. Τώρα, η ηλεκτρική προώθηση η υβριδική καταρχάς μεικτή αλλά στη συνέχεια αμυγός ηλεκτρικ... ηλεκτροκίνηση των αεροσκαφών θα είναι στόχος της δεύτερης γενιάς στο πρόγραμμα Καθαρός Ουρανός. Σίγουρα αυτό παίρνει πάρα πολλά χρόνια να γίνει, αλλά σας είπα ότι γενικότερα η αεροπορία είναι ένας κλάδος με βάθος χρόνου, με χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο και πρέπει να ξεκινάει πράγματα για να μπορέσουν αυτά να καταλήξουν μετά από μία ή δύο δεκαετίες. Ε, μπορούμε λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε τη δουλειά πάνω σε αυτό το στόχο. Ε, αποτελεί αυτό μια δράση επιστημονικά συνεπή. Σε κάθε περίπτωση ο εξυγχρονισμός του κλάδου αυτού είναι πολύ σημαντικός. Η ασφάλεια στις εναερίες μεταφορές ανάγκασαν αυτό το κλάδο να οργανωθεί καλύτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. Έχουμε διάφορες πλατφόρμες ε, πάνω στις οποίες αναλαμβάνουμε κοινή δράση, δεσμευτική δράση. Ο Διεθνής ε, Οργανισμός ε, Πολιτικής Αεροπορίας θα εκδώσει κανονισμό για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όπως επιβάλλει και περιορισμού σε σχέση με τα επίπεδα θορύβου και η χώρη ύπαρσης. Έχουμε λοιπόν τις απαραίτητε βάσεις για να προχωρήσουμε και νομίζω ότι η βούληση είναι κοινή από όλα τα μέρη. Η Ευρώπη δραστηριοποιείται σε αυτό το τομέα, αλλά δεν είμαστε μόνοι και στη ΣΥΠΑ υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα με το πρόγραμμα Clean Sky, καθαρός ουρανός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την τρίτη παρουσίαση αυτή και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στις ερωτήσεις, στις ε, παρεμβάσεις των ε, βουλευτών. Η Καρή Μαντέλη πρώτη. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Εγώ έχω διάφορες ερωτήσεις. Εκ μέρους, ε, μάλλον, προς, την, προς τον εκπρόσωπο των αυτοκινηστών και κάποιες ερωτήσεις για τα των αερομεταφορών. Κάποιος προηγούμενος ε, ομιλητής είπε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αν και το βλέπουμε αρκετά σκούρο το μέλλον. Έχουμε μεγέθη. 40 εκατομμύρια πολίτες εκτίθενται σε, σε ε, εκπομπές ε, και σε μικροσωματίδια PM10 δηλαδή τύπου πολύ αυξημένα κατά 40% από τα επιτρεπόμενα όρια, 400.000 ε, πρόβλη θάνατοι, όλα αυτά λόγω των μικρών σωματιδίων. Και απλώς για να πω δηλαδή, και βλέπω ότι είστε όλοι εδώ, καλό είναι αυτό, 767 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εκτίμηση του κόστους για τη δημόσια υγεία. για να πούμε και ένα μέγεθο. Πώς λοιπόν ο κλάδος των κατασκευαστών αυτοκινήτων δεν μπορεί να σεβαστεί τα 80 μικρογραμμάρια ένα χιλιόμετρο, ενώ σε άλλες χώρες αυτό γίνεται σεβαστό. Εσείς συνδέετε τα όρια με την ταχύτητα. Για την ταχύτητα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, μάλλον από το 2014, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και σοβαρούς δραματισμούς και ως εισηγήτρια της αστικής κινητικότητας μπορώ να σας πω ότι δεν βοηθάτε γιατί αντί να περιορίσετε την ε, τελική ταχύτητα κάνετε τα πάντα <clears throat> ώστε να αποφεύγονται αυτές οι ερωτήσεις να τίθενται παρότι είναι σημαντικές. Άλλο ένα θέμα. Μιλάτε για τεχνολογία. Θυμίζω ότι στην Επιτροπή αυτή δεν υπάρχει καθαρό ντίζελ. Σήμερα μιλάμε για νέα φίλτρα σωματιδίων αλλά με τα φίλτρα σωματιδίων βγαίνουν ακόμη πιο μικρά τα σωματίδια σε διάμετρο από το φίλτρο και δηλαδή είναι ακόμα πιο επικίνδυνα. Επομένως ερώτηση κύριε εκπρόσωπε του κλάδου των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Πότε πραγματικά σκέφτεστε να μετατραπεί ο κλάδος για να εξαφανιστεί ο κινητήρας diesel. Γιατί αν δεν γίνει αυτό σταδιακά θα είναι οι εργαζόμενοι που θα την πληρώσουν χάνοντας τη δουλειά τους. Και θα τελειώσω εδώ, Πρόεδρε, με μία ακόμα ερώτηση για τις Το Τομέας όπου η συσχέτιση με τα, του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι όλο και πιο ουσιαστική. Μιλάμε για τον δίζελ. Μήπως αύριο θα πρέπει να μιλούμε για την ε, σωστή φορολόγηση της κυροζήνης. Γιατί αυτός ο κλίδος ο κλάδο ρηπαίνει και αυτό, όπω πολλοί άλλοι. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, η Μαρία Κίλωνα. Thank you, Chair. Thanks for Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του ομιλητέ. Να θέσω κάποια φλέγοντα ζητήματα για τον κ. Πεντρό. λέει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Αυτοκινήτων, γιατί θεωρώ ότι είπατε ότι δεν πειράζει τόσο πολύ τι γίνεται με τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Γιατί είμαστε άλλωστε μικρός πληθυσμός. Αλλά κοιτώντα ε, τα δικά σας έγγραφα για τη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων στον κόσμο, έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κάνει μεγάλη διαφορά από ό,τι κάνουμε στην Ευρώπη. Τεράστιος ο όγκος αυτοκινήτων αρχή. Ελπίζω λοιπόν να μην μας υποτιμάτε σε καμία περίπτωση και εμάς και την επιρροή μας. Two or three times more car. Γιατί έχουμε διπλάσια και τριπλάσια αυτοκίνητα ποσοστία και αναλογικά. Ακόμα και σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και αυτό φυσικά με ό,τι συνέπειες έχει και για τη ρήπανση και για τα κλιματικά. Ό,τι καλύτερα λοιπόν σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η Στέλλα. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία ερώτηση για ένα πρόσωπο των κατασκευαστών αυτοκινήτων και μία για τον εκπρόσωπο του Clean Sky. Οι κατασκευαστές φορτηγών ή τέλο αυτοκινήτων λένε ότι μπορούμε να τους εμπιστευτούμε για την εξοικονόμηση καυσίμου. Παράλληλα υπάρχουν κατηγορίες για παράνομη ρύθμιση τιμών μεταξύ του 97 και του 2011 ότι έχουν συμφωνήσει δηλαδή τις τιμές με την εισαγωγή πράσινης τεχνολογίας. Επομένως, με αυτό το δεδομένο, γιατί να σας εμπιστευτούμε. Δεύτερη ερώτηση. Για τις αεραμεταφορές. Στις διαφάνειες είδα συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και διαρωτώ με κατά πόσον Αυτό ήταν οι εκπομπές συνολικής ανάπτυξης ή το δυναμικό, οι προβολές ανάπτυξης. Αλλά παράλληλα πρέπει να προσθέσει κανείς σε ποιο ύψος εκπέμπονται αυτά. Γιατί έχουν διαφορετικό αντίκτυπο. Ευχαριστώ κύριε Σπίπερ. Νομίζω ότι βασικά πήρα το λόγο για να σχολιάσω αυτό που είπε ο συνάδελφο, αγαπητοί συνάδελφοι, από την αριστερά. 12 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται με όλε τι οικογένειε του στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Το συνειδητοποιείτε αυτό. Συνειδητοποιείτε ότι 75% ενό αυτοκινήτου μικρομεσαίων επιχειρήσεων παράγεται από μικρομεσαίε επιχειρήσει, με λιγότερα από 200 ε, εργαζόμενους και ότι όλα αυτά τα σενάρια για την απαγόρευση τέτοιων τεχνολογιών τι σημαίνει. Ανησυχώ, ανησυχώ πάρα πολύ. Μήπως ξεκινάμε μια επιχειρηματολογία υπερβολικά μονόπλευρη. Φυσικά υπήρξαν ε, τα σκάνδαλα και φυσικά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πέτοι. Αλλά δεν είναι αυτό που αφορά όλη την αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία κλίκα, αν θέλετε, εγκληματιών. Αλλά για να κατηγορήσουμε και να καταδικάσουμε όλη την αυτήν αυτοκινητοβιομηχανία πιστεύω ότι είναι λάθος και θα ήθελα να το διευκρινίσω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ζήτησα και εγώ το λόγο, γιατί ζήτησα και το λόγο. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε μονόπλευροι σε μια δημοκρατία. Στην αυτοκινητοβιομηχανία θέσαμε τα eco-liner, αυτά τα τεράστια φορτηγά, και υπάρχουν ε, και έρευνες που καταδεικνύουν ότι το 35% ε, μπορεί να γίνει, τα μεταφορών μπορεί να γίνει συνδρομικά και ένα άλλο μεγάλο ποσοστό μπορεί να γίνει οδικά. Ε, γενικά ο αντίκτυπος δεν είναι θετικός. Και δεύτερο σημείο, και στα αυτοκίνητα έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια. Μας τα είπατε, όντως. Αλλά ο συνολικός απολογισμός δεν είναι καλύτερος γιατί τα αυτοκίνητα είναι πιο μεγάλα, πιο βαριά και είναι και πιο πολλά. Άρα καταναλώνουν πιο πολύ. Τα SUV λοιπόν αυξήθηκαν στη χρήση του και είναι πολύ πιο βαριά στη χρήση και στην κατανάλωση από ότι άλλα αυτοκίνητα. Και εδώ λοιπόν πρέπει να αναφερθούμε σε ό,τι αφορά την ε, ναυτιλία. Η ναυτιλία χρησιμοποιεί και τα μεγάλα πλοία χρησιμοποιούν αργό πετρέλαιο. Αυτό αποτελεί ε, προϊόν της πετρελαιοβιομηχανίας. Γιατί δεν ε, απαγορεύεται λοιπόν ε, αυτό το καύσιμο του οποίου η καύση είναι τόσο επιβλαβής. Με κανονικό ντίζελ θα είχαμε καλύτερες, καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι με το πετρέλαιο. Και οι αεροπορικέ μεταφορέ αυξάνονται μέσω των επιδοτήσεων, μια και δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν φόρο επιτικής κυριοσύνη κτλ. Αλλά φυσικά είναι υπέρ των ε, μειώσεων και στην ε, αεροπορική μεταφορία. Αλλά το γεγονό ότι μεταξύ ε, Φραγκφούρτη και Στουτγκάρδη κάθε χρόνο έχουμε τόσε πολλέ πτήσει. θεωρώ ότι είναι παραλογισμό Βερολίνο, Ανόβερο, Παρίσι, Βρυξέλλε. Ε, εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν πλέον πτήσει. όχι τόσες πολλές τέλο πάντων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε σε ό,τι αφορά το όριο ταχύτητας. Στη Γερμανία δεν είναι η μοναδική χώρα που δεν υπάρχει τέτοια πτυχή ε, περιορισμός. Ακόμα και στη ΣΥΠΑ, πρακτικά είναι 120-130 χιλιόμετρα ανά ώρα το όριο αυτό. Για την Γερμανία, λοιπόν, χρειαζόμαστε μέτρα ερευνών. Πρέπει δηλαδή τα αυτοκίνητα να οδηγούν 200-250 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, για τη Γερμανία μιλάω. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκέ δοκιμέ για όλου ε, ίδιε. Αν μόνο στη Γερμανία έχουμε αυτοκίνητα που τρέχουν με 250 χιλιόμετρα, μήπω χρειάζονται πιο αυστηρά μέτρα. Και τελευταίο, και τελευταίο ζήτημα και με αφήνει να ολοκληρώσω και ο κύριος Πίπερς, μεγάλη μου τιμή. Στην ερώτησή σας θα ήθελα να επανέλθω επειδή σα ακούω. Η αυτοκινητοβιομηχανία με τις ε, θέσεις Σωστό αυτό. Έτσι αρτρώεται. Έξυπνος, αλλά πολύ πριν από την εποχή του τότε είχε αναμορφώσει πριν από 10 χρόνια την Diamond Chrysler και είχε δηλώσει ότι ως αυτοκίνητο βιομηχανίας έχουμε μέλλον μόνο αν καταστούμε όμιλος ε, κινητικότητας. Ε, έφτιαξαν λοιπόν ε, αυτοκινητοδρόμους, φορτηγά, ECA και ακόμα και ποδήλατα. Και ο κ. Φρέμπτ τα πούλησε όλα και σήμερα η Daimler εξαρτάται μόνο από της πώληση αυτοκινήτων. Αν υπήρχε μια γενικότερη όμως τέτοια, ένα γενικότερο σχέδιο, θα μπορούσε να υπήρξε, να υπάρξει κατάσταση των θέσεων εργασία αυτή και παράλληλα να προστατεύεται το περιβάλλον. Αυτό είναι το μέλλον τη αυτοκινητοβιομηχανία. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι θα επιβιώσουν και θα έχουν μέλλον μόνο εκείνοι οι όμιλοι οι οποίοι θα έχουν ένα μελλοντικό συνολικό σχέδιο για όλη την κινητικότητα. Δυστυχώ όμω πλέον για την Daimler Chrysler είναι αργά. Νομίζω ότι εσεί που οδηγάτε και Mercedes έχετε πιο πολλέ εμπειρίε από ότι εγώ. Το λόγο τώρα έχει ο Ιβο Μπελέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω μία ερώτηση στα Ολλανδικά προ τον κύριο Χιούτζα ε, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, γιατί είμαστε στα πρόθυρα, είμαστε μάλλον πριν από την 25η διάσκεψη των μερών στο Παρίσι και ξέρουμε ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια από όλους τους τομείς και όλοι προσβλέπουμε στη συμφωνία όχι μόνο στον ΙΚΑΟ και στον ΑΕΜΟ για τη συμφωνία που θα πρέπει να συναυτεί πριν τέλη το επόμενο έτος για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πείτε μας λοιπόν ποιες είναι οι προβλέψεις, οι προπτικές για την επίτευξη μια τέτοια συμφωνία πριν τα τέλη του επόμενου έτου. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να σα υποδείξω και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που θα παρουσιαστεί αύριο το πρωί στο Κοινοβούλιο για τις εκπομπές της Διεθνούς Αεροπορίας και της Ναυσιπλοείας. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και πολύ ανησυχητικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αυτές, αν δεν καταφέρουμε να μειώσουμε δραστικά αυτές τις εκπομπές. Δεν φτάνει λοιπόν μέχρι το 2020 να προσπαθήσουμε απλά να ελέγξουμε τις εκπομπές. Θα πρέπει δραστικά να τις μειώσουμε. Γιατί η δάλος, το ποσοστό της ναυσιβλογίας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθεί δραματικά. Είναι ναυσιπλοεία δηλαδή καταβάλει πολύ λιγότερες προσπάθειες ενώ στους υπόλοιπους τομείς γίνεται πιο μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις λοιπόν ακούσατε και έχετε τη δυνατότητα τώρα να απαντήσετε με την ίδια σειρά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους από δεξιά προς τα αριστερά. Έχω υπάρξει διπλωμάτη στο παρελθόν και αυτό βοηθάει σήμερα. Τώρα, ως προς τα σωματίδια να σας πω ότι πολλές είναι οι μελέτες που δίνουν πολλά διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία και πολλά και διαφορετικά συμπεράσματα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει μια καλή μελέτη που να λέει αυτή είναι συγκεκριμένα η συμβολή των επιβατικών οχημάτων, ε, ε, φορτηγών ή αυτή είναι η συμβολή της θέρμασης. Τα βάζουν όλα στο ίδιο καλάθι και ειδικά ως προς το Γιατί να ευθύνεται το ντίζελ σήμερα που αυτή τη στιγμή το υφιστάμενο πρότυπο είναι μηδέν στο δίζελ. Σε μια, στη μέση κατάσταση ένα δεκαετές αυτοκίνητο πράγματι ένα αυτοκίνητο δεκαετών εκπέμπει πολύ. Όλοι το γνωρίζουμε. Αν πάτε όμως σε μια αντιπροσωπεία και ζητήσετε ε, το, το δίζελ με το υψηλότερο στάνταρ έχει μηδέν εκπομπή σωματιδίων και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη τα τελευταία 20 και 30 χρόνια. Λέγαμε ναι, είναι καλό το ντίζελ γιατί έχει πολύ χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και όλες οι πολιτικές πάνω στις οποίες ε, συμφωνούσαμε όλοι από κοινού είχαν στο επίκεντρο το διοξιδίο του άνθρακα και γι' αυτό υπήρξε και συγκεκριμένη τεχνολογία για το διοξίδιο του άνθρακα. Μπορεί να συζητήσει κατά πόσο θα κάνει μεταστροφή προς άλλες τεχνολογίες για να ε, φτάσει σε ένα σημείο ισορροπίας. Αλλά γι' αυτό είχαμε τα Euro Standard από το 1 μέχρι το 6 που ισχύει σήμερα το το 6. Αυτή ήταν η πολιτική μας και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς. Τώρα, ως προς το... την κατάσταση στην Ευρώπη. Απαντώ ναι. Μάλλον εμείς έχουμε το ε, περισσότερο στόλο αυτοκινήτων, αλλά έχουμε και το πιο αυστηρό στόχο. Αν δείτε την Κίνα, για παράδειγμα, ή την Κορία, περιμένουν αυτοί να δουν τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι και μετά ακολουθούν. Το στάνταρ το 95, το Euro 95, είναι και το πιο αυστηρό στον κόσμο. Νομίζω ότι ε, δείχνουμε τη σοβαρότητά μας και είμαστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Εάν δούμε τι συμβαίνει στην κινέζικη αγορά, η οποία μάλλον σε ένα-δύο χρόνια θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στην Ευρώπη, θα είναι διπλάσια ηλικία του μέσου αυτοκινητού, άρα τα αυτοκίνητα θα έχουν παραχθεί στη δεκαετία του 80, φανταστείτε τις επιδόσεις τους και μιλούμε για εκατομμύρια οχήματα ε, τα οποία ε, θα κυκλοφορούν, θα εκπέμπουν αέρια τα οποία ταξιδεύουν, δεν μένουν στο δύο μέρος και φτάνουν τελικά στην Ευρώπη ούτως ή άλλως ο κύκλος ζωής, ο οικονομικός και η πραγματικότητα στον πλανήτη είναι διαφορετική και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όλα αυτά. Τώρα, αν διεράσω, διαιρέσω αυτό το δωμάτιο σε μισά, σε δύο ίσα τμήματα, σίγουρα το πρώτο δεν θα με εμπιστευτεί και το δεύτερο ε, θα με εμπιστευτεί για το μέλλον. Κάθε φορά ε, υπάρχουν αρνητικές αντιδράσεις. Στις περιπτώσεις καρτέλ ε, φορτηγών ή άλλες περιπτώσεις με εξαπατήσεις, να σας πω ότι καμία δεν αποδείχθηκε και σε καμία δεν συμφώνησε το δικαστήριο. Τώρα το να μας αρέσει να μας αρέσει είναι άλλο θέμα. Όμως υπήρξαν υποθέσεις που ε, έτυχαν αντιμετώπισης, υπήρξαν αποφάσεις και βεβαίως συμφωνούμε ότι ναι, <clears throat> όποιος παραβαίνει ε, τους κανόνες θα πρέπει να τιμωρείται και θα τιμωρηθεί. Έρχομαι τώρα στα σχόλια του Προέδρου ως προς τα πολύ μεγάλα φορτηγά, τα mega αλλά και τα επιβατικά οχήματα. Ναι, όλοι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Τα mega trucks μπορεί να μας βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα, μπορεί να είναι πολύ καλά σε ορισμένες χώρες γιατί βελτιώνουν τις επιδόσεις και παράγματι βελτιώνουν, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση διοξιδίου του άνθρακα με τα mega trucks, τα mega φορτηγά, όμως σε κάποιους δεν αρέσουν και είναι δημοκρατική η συζήτηση, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω έτσι όπως έγιναν οι ερωτήσεις. Για τα καύσιμα της ναυτιλίας, ε, εντός του Marplan 6 που ανέφερα νωρίτερα, υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την ε, περιεκτικότητα βαρύτερου καύσιμου που θα περιοριστεί από 3,5% στο 0,5% μέχρι το 2020 κατόπιν επανεξέτασης, γιατί μιλάμε για 200 εκατομμύρια πρόσθετου καυσίμου, τόνους πρόσθετου καυσίμου, πρέπει να δούμε και τη διαθεσιμότητά του. Εφόσον όμως αποφασίσουν τα μέρη, στο παράδειγμα 6, ότι δεν υπάρχει το επαρκές καύσιμο, θα μετακινηθεί ο στόχος το 25, το 2025. Πάντως αυτό το, αυτή η διάταξη θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Τώρα, δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας για τις ε, διατάξεις ε, της Διεθνούς Συμφωνίας στην COP21 αναφερθήκατε σε κάποια άλλη διεθνή συμφωνία, στο τι κάνει ο IMO. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για την αύξηση των ε, εκπομπών της ναυτιλίας. Ναι, αυξάνονται οι εκπομπές. Και τοποθετούνται μεταξύ του 50 και του 250% μέχρι το 2050 όπως έλεγα. Αλλά ανασκάφος το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη σύγκριση με άλλους κλάδους, έχουμε εισαγάγει υποχρεωτικές διατάξεις ε, ενεργειακής απόδοσης για το κάθε σκάφος. Όμως, εφόσον αυξάνεται και μεγεθύνεται το παγκοσμίο εμπόριο και ο όγκος των εμπορευμάτων και παρακολουθεί η ναυτιλία τις απαιτήσει αυτές, τότε θα αυξάνονται και εκπομπές, διότι ακόμα και αν μειώσεις τις εκπομπές κάθε σκάφους, συνολικά θα αυξάνονται οι εκπομπές. Υπάρχει λοιπόν πρόκληση και είναι πρόκληση για όλους. Γιατί έχουμε την παγκόσμια ζήτηση και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο. 171 μέλη όπως σας έλεγα έχουμε. Μεταξύ των οποίων χώρες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ στην ανάπτυξη της δική τους, ε, του δικού τους μερίσματος στο παγκόσμιο εμπόριο. Επομένως χρειαζόμαστε ισορροπία μεταξύ της μείωση των εκπομπών αυτού του τομέα και της ε, υπηρέτησης της παγκόσμιας οικονομίας και του εμπορίου. Και αυτό είναι θέμα και για τους ε, πολιτικούς ηθήνατους παντού στον κόσμο. Τώρα, ή στο πλαίσιο του IMO έχουμε βελτιώσει όλα τα πρότυπα σχεδιασμού και να στους σκαφών, τα συστήματα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση σκαφών και είχαμε και πρόσφατες συνεδριέσεις επ' αυτού, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μέτρα κατάλληλα για τον παγκόσμιο στόλο. Και συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή. Γνωρίζοντας το τι συμβαίνει. Απλώς δεν ήμουν βέβαιος για την ερώτησή σας επί των διατάξεων, αν θέλετε να διευθυνίσετε. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Και θα το πω στα αγγλικά και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου υπάρχουν σαφέστατα αιτήματα προς τον ΚΑΟ και τον IMO για να επιτευχθεί μια διεθνή συμφωνία εντός του IMO μέχρι το τέλος του 2016 εκ μέρους της COP21. Δηλαδή τι θα κάνει ο IMO προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία μέχρι το τέλος του 2016. Γιατί υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κάποια προβλεψιμότητα σχετικά με την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ για τη διαφήμιση, λέει ο Μελτής Στον IMO εξετάζουμε περαιτέρω μέτρα εδώ και αρκετά χρόνια. Από το 2003 <clears throat> είχαμε ε, μέτρα της αγοράς ε, που εξετάζαμε την εφαρμογή τους, αλλά το θέμα είναι το παγκόσμιο πλαίσιο, το εθνές πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Προφανώς εργαζόμαστε υπό το πρωτόκολλο του Κιώτο, όπου υπάρχουν και οι χώρες παρετήματος 1, για τη συνεργασία με τον ΙΚΑΟ και τον ΑΕΜΟ, και είναι θεμελιώδη ζήτημα για τον ΑΕΜΟ αυτό. Γιατί όπως σας είπα ρυθμίζουμε τα τυναφιλία, τα σκάφη και αυτό υπό κάποια έννοια προσπαθεί να αντισταθμίσει την αρχή αυτή με την αρχή της διαφοροποιημένης ευθύνης που βλέπουμε υπό το UNCCC. Τώρα, πολλά εξαρτώνται από το τι θα τεθεί στο, στο Παρίσι και όπως και εσείς ενδιαφέρομαστε πάρα πολύ να δούμε το το αποτέλεσμα και ευχόμαστε να είναι επιτυχίες αποτέλεσμα. Το οποίο θα θέσει το πλαίσιο για το πού θα πάμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το, η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει με την ενδεχόμενη φορολόγηση της κυροζήνης. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που του σηκώνεται το μαλλί όρθιο όταν ακούνε για φόρους. Γιατί όχι, απαντώ. Με ένας φόρος στην κυροζήνη θα αυξήσει λίγο την τιμή της αεροπορικής μεταφοράς και τίποτα άλλο. Η εναλλακτική είναι τα βιοκαύσιμα, τα οποία δεν έχουν οριμάσει για να χρησιμοποιηθούν βιομηχανικά στην αεροπορία, στη βιομηχανία, αλλά πάνω σε αυτό δουλεύουμε. η αεροπορία άλλωστε θα είναι περιθωριακός χρήστης των βιοκαυσίμων. Είναι όμως σημαντικό για την ίδια. Υπάρχουν όμως και άλλες τεχνολογίες και υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που ήδη χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και που χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, η εν μέρη τουλάχιστον μετάβαση στα βιοκαύσιμα είναι ένας από τους απαραίτητους, ε, ένα από τα απαραίτητα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους το 2050. Τώρα, αν κάποια στιγμή αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμο να, περάσει, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέσω της φορολόγησης της κυροζήνης, ε, γιατί όχι, απαντώ. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια διαφορετική οδό που είναι το σύστημα εμπορίας ρήπων που εφαρμόζονται στην αεροπορία. Έχει υποστεί ε, κάποιες ε, μεταλλάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και αναταραχές τις γνωρίζετε. Οι αερομεταφορές και η αεροναυπηγική πράγματι είναι απολύτως παγκοσμιοποιημένοι κλάδη στην οικονομία και θα πρέπει κανείς να το προσέχει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η Ευρώπη να ε, μη βρίσκεται στην, πρωτοπορία ως προς τη λήψη νέων μέτρων, σαφώς και θα πρέπει να βρίσκεται, αλλά δεν είναι μόνη της. Και σε επίπεδο ΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και σε επίπεδο άλλων οργανισμών οργανώνεται αυτός ο κλάδος και από εκεί περνάει, από, από αυτούς τους αγωγούς περνάει η έβρεση κοινών ε, λύσεων. Ο ΙΚΑΟ ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας εργάζεται εντατικά για τη θέσπιση ενός κανονισμού προτύπων και στάνταρ ε, ορίων για το διοξίδιο του άνθρακα που θα είναι τόσο αυστηρή όσο και τα όρια που έχει θέσει για την ηχορύπανση που τα αναθεωρεί ο ΙΚΑΟ σε τακτά χρονικά διαστήματα, την παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας και εκπροσώπων των κρατών. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα υπάρξει κανονισμός από πλευρά ΙΚΑΟ. Δεν θα σας δώσω αριθμητικά στοιχεία σήμερα, όμως η βάση είναι ευρεία πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε ώστε ο ΙΚΑΟ να θέσει στόχο που να είναι εφικτός αλλά και επαρκώς φιλόδοξος συνάμα. Και όπως συνέβη και με την ηχώρη ύπανση, θα πρέπει και στο διοξίδιο του άνθρακα να ε, συνοδευτούμε ε, σε αυτή την πορεία από τις τεχνολογικές εξελίξεις ε, προκειμένου να φτάσουμε σε στόχους εφικτούς και όχι τελείως μη προσβάσιμους. Τώρα, Βρυξέλλες Παρίσι, Παρίσι Μασαλία, ε, Βρυξέλλες Περπινιάν. Ευχαρίστως να πάω με το τρένο. Δεν ε, είναι απαραίτητο να ε, υπάρξει λόμπι αεροπορίας ως προς αυτό. Είναι θέμα βέλτιστης χρήσης και βέλτιστης επιλογής μεταφορικού μέσου. Αν η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύξει ε, μέσω συντροδρομικής ε, μεταφοράς πιο αποτελεσματικό από την αέρια μεταφορά, έχει καλός. Μιλούμε για διατροπικές μεταφορές. Είναι θέματα που συζητούνται σε εθνικό, σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το βασικό σε σχέση με την ανάπτυξη των αέριων μεταφορών, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τη μεταφορά από τη μία πόλη στην άλλη της Ευρώπης. Έχει να κάνει με τη μεταφορά από και προς την Ασία, από και προς τις αναδυόμενες ή άρτη αναδυθήσεις χώρες. Ε, με τη μεταφορά από και προς τη Μέση και από Ανατολή. Άρα ε, το διακύβευμα είναι απολύτως παγκόσμιο για άλλη μια φορά. Και τέλος, μου τέθηκε μία ερώτηση για τη φύση των αριθμητικών στοιχείων. Ε, δεν μιλούμε για αριθμητικά στοιχεία, μιλούμε κυρίως για ε, τάσεις. Ναι, είναι οι εκπομπές ε, οι ακαθάριστες αν θέλετε και μετά υπάρχει επιστημονική επεξεργασία των επιστημονικών δεδομένων και αριθμητικών στοιχείων για να δούμε πώς ακριβώς αυτές πλήττουν το κλίμα αναλόγως με το υψόμετρο και το καθεξής. Σε κάθε περίπτωση οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τη μείωση των εκπομπών πρέπει να είναι αναλογικές ανεξάρτητα με το πραγματικό ποσοστό, το κατόφλι αν θα το θέσουμε στο 3, στο 4, στο 5%. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν... Α, υπάρχει άλλη μια μικρή ερώτηση. Μία μικρή επερώτηση για τον κύριο από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πείτε μας, μία μάρκα αυτοκινήτων diesel που δεν έχει εκπομπές ε, σωματιδίων. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Νομίζω ότι ο κανονισμός ε, ορίζει σαφώς τι πρέπει να ισχύει και όλοι ακολουθούμε αυτές τις κανονισμούς. Όλα τα μέλη μας νομίζω είναι στα νόμιμα όρια και πληρούν τους νόμιμους όρους. Μάλιστα. Και η έλλειψη απάντηση αποτελεί απάντηση. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις και για τις ερωταπαντήσεις. Ε, νομίζω ότι σε ένα πράγμα είμαστε όλοι σύμφωνοι. Θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε όλους τους τομείς. Δεν ξέρω κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή, μετατόπιση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό που θα είναι καθαριστικό και τα ακούσαμε πολλές φορές είναι ο καθολικός και παγκόσμιος χαρακτήρας. Στις ΕΙΠΑ, για παράδειγμα, έχουμε 800 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Όποιοι δηλαδή μπορούν και έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, έχουν στατιστικά αυτοκίνητα, ακόμα και αν κάποιε οικογένειε έχουν πολλά αυτοκίνητα και κάποιε άλλε δεν έχουν αυτοκίνητα, και στην Κίνα είναι 40 το αντίστοιχο το, το αντίστοιχο αριθμό αυτοκινητών. Αλλά δεν μπορούμε κι εμεί ε, με τι με τι Mercedes και τι Peugeot να πάμε στην Κίνα και να πούμε ότι κοιτάξτε να μην οδηγείτε γιατί είναι επικίνδυνη η οδήγηση. Όχι, μπορούμε να ακολουθήσουμε απλά και να δώσουμε το καλό παράδειγμα και εδώ η Ευρώπη είναι global player, είναι παγκόσμιος φορέα. Θα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την κινητικότητα και να προστατεύσουμε το κλίμα. Αλλά να το δείξουμε, όχι απλά να μιλάμε. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Και εγώ ως Γερμανός θυμάμαι και την ε, κατηγορηματική επιτακτική ανάγκη να ζει κανείς με τον τρόπο με τον τρόπο που είναι δυνατό να ζήσει κάθε άνθρωπο στον κόσμο, όχι μόνο κάθε άνθρωπο στον δυτικό κόσμο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς είναι ο κόσμος, όχι μόνο πώς είναι ο κόσμος εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε και την παγκόσμια προοπτική υπόψη. Πολλά μπορούμε να πετύχουμε και χρειάζεται λοιπόν δίκαιος ανταγωνισμός. Οι 300 πτήσεις μεταξύ Στουτγκάρτης και Φραγκφούρτης, ε, κοιτάξτε, είναι καλή η, η σύνδεση η συνδρομική που υπάρχει, μόνο που είναι διπλάσια στη τιμή. Χρειάζεται λοιπόν τέτοιο ανταγωνισμό. Είτε να πληρώνουμε όλοι οι ΦΠΑ είτε όχι. Πολλά λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά θα συζητηθούν στο Παρίσι και ακριβώς λόγω και εν του Παρισιού κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι όλοι πήραν το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και έτσι ολοκληρώνω τη σημερινή μας εκδήλωση και στο τέλος της συνεδρίασης ε, της Επιτροπής Μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.